Ladies and gentlemen, Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καθίστε. Θα αρχίσουμε αμέσως. Thank you. Welcome to the... Καλώς ήρθατε λοιπόν στη συνεδρίαση της υποεπιτροπής μας. Καλώς ορίζω τα μέλη, τους καλεσμένους και τους παρατηρητές. Όπως ε, συνήθως έχουμε μετάφραση και διερμηνία για, τις, ε, για τα τακτικά μέλη της Υποεπιτροπής της Ασφάλειας και Άμυνας και επίσης υπάρχει ε, μετάδοση απευθείας από το διαδίκτυο. Περνάμε κατευθείαν στην ημερήσια μας διάταξη. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και ιδιαιτέρως μετά τον βομβαρδισμό της Μαριούπολης στην Ανατολική Ουκρανία αποφάσισα να συμπεριλάβω στην ημερήσια διάταξη ένα σημείο για σύντομη ενημέρωση για το θέμα αυτό που εντάσσεται στην εντολή της Υποεπιτροπής μας και θα επικεντρωθούμε σε πολιτικά και στρατιωτικά σκέλη της κατάστασης αυτής και η ενημέρωση θα γίνει από τον πρέσβη Ήλις Κωνσταντίνη Λισέεφ που είναι μόνιμος ε, αντιπρόσωπος της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν συμφωνείτε λοιπόν αυτή την αλλαγή, την προσθήκη στην ε, ημερήσια μας διάταξη, θα ακούσουμε αυτή την ενημέρωση αμέσως μετά την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε για την Βοσνία και Ριζεγοβίνη. Ωραία, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, άρα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη και επιτρέψτε μου να καλωσορίσω θερμότατα το πρώτο και επιφανή καλεσμένο μας, τον στρατηγό Έντριαν Μπράτσο, που είναι καταπληκτικός ε, διοικητής και αυτή τη στιγμή υποδιοικητής της Ανωτέρας Συμμαχικής Διοικήσεως Ευρώπης ε, και της επιχείρησης Αλτέα στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Η πείρα του είναι τόσο πλούσια που καλύτερα να μην χρονοτριβούμε άλλο και να του δώσω κατευθείαν το λόγο για να μας κάνει την ενημέρωση. Είχε εμπειρία στα νησιά Φόλκλαντ, στο Αφγανιστάν και στα Δυτικά Βαλκάνια. Πλούσια πείρα στρατιωτική. Σας απευθύνω λοιπόν εγκάρδιο καλωσόρισμα στρατηγέ μου και θα ακούσουμε την ομιλία σας προς την Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για τα ευγενικά σας λόγια. Αγαπητοί εξάτιμοι ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία αυτή για πρώτη φορά να έρθω στην Επιτροπή σας υπό το ρόλο μου του υποδιοικητή της Ανωτέρας Συμμαχικής Διοίκησης Ευρώπης στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Ε, συμμετείχα ως διοικητής ε, ενός τάγματος ε, στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, στην ΕΣΦΟΡ και είδα ειδήσόμαση την προσπάθεια, τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι λαοί μας να αποκαταστήσουν την ειρήνη στα Δυτικά Βαλκάνια. Και χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί από την εποχή της Έσφορ βλέπω σημαντική διαφορά και πρόοδο. Παρόλο που πολιτική κατάσταση δεν είναι το βασικό μέρημά μου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για αυτά τα θέματα. Η πολιτική στη Βοσνία Ζεγοβίνη φαίνεται ότι έχει εγκλωβιστεί σε μία αποτελμάτωση μετά τη συμφωνία των Dayton και είναι δύσκολο να ληφθούν αποφάσει και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική διακυβέρνηση. Αυτό επηρέασε και την κατάσταση τη Άμυνα και ασφάλεια, όπω και όλου του κλάδου διακυβέρνηση στη Βοσνία και Ζεγοβίνη. Και μετά τι περσινέ εκλογέ. Φαίνεται παρόλα αυτά ότι υπάρχουν κάποιοι λόγοι για συγκρατημένη αισιοδοξία και μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία Γερμανίας Ηνωμένου Βασιλείου για να ξαναξεκινήσει η διαδικασία ολοκλήρωση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις για οικονομικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις και κυρίως για τα κοινωνικά θέματα που είναι το άμεσο, ε, η άμεση ανησυχία του πληθυσμού ειδικά μετά τις ε, αναταραχές που είχαμε το περασμένο Φεβρουάριο. <clears throat> Και έχουμε διάφορες πλατφόρμες φετεράνων πολιτικών προκειμένου να, γίνει, να ενεργοποιηθεί πάλι η διαδικασία της ένταξης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχαμε και θετικά σημεία σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για μια ένταξη και στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα ακόμη και το, ο Σέρβος εκπρόσωπος ε, στην Προεδρία τάχθηκε υπέρ της ε, πρόθεσης υποψηφιότητας της Βοσνίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ελπίζουμε βέβαια όλα αυτά τα θετικά σημάδια να ε, μεταφραστούν και σε έμπρακτη δράση που θα είναι πραγματική απόδειξη προόδου στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και μάλιστα ενώ οι εθνικοί θεσμοί είναι σχετικά δύναμοι και αναποτελεσματικοί, τα καλά νέα είναι ότι οι ένοπλε δυνάμει τη Βοσνία και είναι από τα λίγα σώματα που ε, φαίνουν κοντά και σε συνεργασία και τους ανθρώπους και από τις τρεις ε, κοινότητες και πραγματικά είναι ε, το καμάρι της Βοσνίας και Ριζεγοβίνης. Και μάλιστα την πέρυσι ε, ο στρατός αναγνωρίστηκε από τον πληθυσμό γιατί συνέβαλε τα μάλα στην, στις, στις σωστικές ε, ενέργειες ε, στις περσινές πλημμύρες και μάλιστα συμβάλλει στη σταθεροποίηση της κατάστασης ε, και συμμετέχει μάλιστα και σε μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Και ενώ η u παρακολουθεί εκ του και στην κατάσταση της ασφάλειας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, σήμερα η εκπαίδευση και η δημιουργία ικανοτήτων είναι το βασικό μας μέλημα. Και οι σχετικές προσπάθειες ε, χαιρετίστηκαν ε, στη Βοσνία Ριζεγοβίνη, γιατί πραγματικά βελτιώνουν τις ικανότητες ε, της χώρας αυτής. Βέβαια τα πλεονεκτήματα θα παραμείνουν περιορισμένα, δεν σημειωθεί πρόοδο στη μεταρρυθμίση της άμυνας, ώστε και οι άνοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τα εσωτερικά, γραφειοκρατικά και διαφορετικά προβλήματα της χώρας που επηρεάζουν αυτή τη στιγμή και περιορίζουν τις δικές μας προσπάθειες εκπαίδευσης. Και μάλιστα χωρίς ε, μια ένα στρατηγικό όραμα για τις ένοπλες δυνάμεις και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας ε, δύσκολο θα είναι να ληφθούν ε, αποφάσεις για δημόσιες προμήθειες και άλλα θέματα της αμυντικής πολιτικής συνεργαζόμαστε στενά και με το ΝΑΤΟ για να, συνεργάσουμε, για να συνδυάσουμε τις προσπάθειες για δημιουργία ικανότητας και εκπαίδευσης και ενώ το ΝΑΤΟ επικεντρώνεται σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, εμείς προωθούμε ε, την εκπαίδευση. Έχουμε μάλιστα κοινούς στόχους με το ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ συντονίζει διμερείς προσπάθειες και προσφορές για εκπαίδευση. Πέρυσι Όλοι οι δραστηριότητε μα για εκπαίδευση και δημιουργία ικανοτήτων ολοκληρώθηκαν βάσει σχεδίου και συνεχίζεται η πρόοδο σε πολλού τομεί. Συνεργαζόμαστε με τι ένοπλε δυνάμει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ώστε να καταλήξουμε σε ένα κοινό πρόγραμμα εκπαίδευση για ειδικευμένη εκπαίδευση. Και μάλιστα μετά τη βασική εκπαίδευση οι, οι στρατηγικοί απασχολούνται σε φρουρέ, και μάλιστα Έχουμε ειδικά προγράμματα στη, στο διάμεσο κατάστημα μεταξύ των βαρδιών που έχουν, αλλά προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και οι δικοί τους εκπαιδευτές ε, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μάλιστα έχουμε ε, όλο και περισσότερες συλλογικέ εκπαιδεύσεις. Μετά τις πλημμύρες ε, του Μαΐου στη Βοσνία ριζεγοβινη οι βασικές μας ασκήσεις με τις ένοπλες δυνάμεις μεταφράστηκαν σε μια έμπρακτη προσπάθεια διάσωσης προκειμένου να επικεντρωθούμε στον προγραμματισμό και στον έλεγχο και να συνεργαστούμε με τις πολιτικές αρχές. Και με τα τεχνικά εμπόδια και ο στρατός της Βοσνίας Ερζεγοβίνης απέδειξε την αποτελεσματικότητά του και τη δέσμευσή του να βοηθήσει το λαό της Βοσνίας. Σε ό,τι αφορά την, το ρόλο της U4 για τη δημιουργία ενός ε, σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος, με ε, τις ε, περιορισμένες δυνατότητες που έχουμε πια και με την ε, αλλαγή της δομής δεν έχουμε πια πολλές ευκαιρίες και χωρίς ε, ενίσχυση να επέμβουμε στη δημιουργία ασφάλους περιβάλλοντος. Και μάλιστα η διαδηλώσει που έγιναν πριν από ένα χρόνο εξαιτίας της αρέσκειας της οικονομικής παρολίγο να ξεφύγουν από τον έλεγχο. Δημιουργήθηκαν και επεισόδια βίας. Οπότε, ακριβώς επειδή η δυσαρέσκεια ε, εξακολουθεί να υπάρχει και δεν έχει αντιμετωπιστεί ούτε σε επίπεδο κεντρικό, ούτε σε περιφερειακό, ο ε, εξακολουθεί και μάλιστα οι συνέπειες των σοβαρών πλημμυρών του Μαΐου επιδήλωσαν την οικονομική κατάσταση και η αναποτελεσματική κυβερνητική δράση έχει διευρύνει το φάσμα μεταξύ των πολιτικών και το χάσμα μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών. Και παρόλο που έγιναν κάποιες βελτιώσεις στο συντονισμό και στην αμοιβαία στήριξη μεταξύ των, ε, αστυνομικών δυνάμεων των καρτονιών, ε, η αστυνομία ε, δεν μπορεί να επέμβει αποτελεσματικά σε περίπτωση που οι διαδηλώσεις αποκτούν ένα βίο χαρακτήρα. Και από τη που δεν θα έχουμε πραγματική πολιτική πρόοδο, η δυσαρέσκεια του κοινού που δημιουργεί αστάθεια παραμένει ε, ζωντανή και δημιουργεί κίνδυνο. Οπότε υπάρχει ε, αυτός ο κίνδυνος ε, για μια έξαρση της βίας, γιατί η πολιτική δυστυχώς για να, εξασφαλίσουν την υποστήριξη επικεντρώνονται σε ίσονο σημασία θέματα. Βέβαια η U4 συμβάλλει σημαντικά στο θέμα της διαχείρισης των πλεονασμάτων, των πυρομαχικών και των εκρηκτικών. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό, ώστε να εξασφαλίσουμε ασφαλέστερο και πιο προστατευμένο περιβάλλον στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη καταρχήν και δεύτερον να αποφύγουμε την διαρροή πυρομαχικών και όπλων προς τις περιοχές όπως ε, Λιβύη, Συρία, Ιράκ ή σε ευρωπαϊκές χώρες γιατί κάποια τέτοια πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν ε, πρόσφατα στις επιθέσεις στο Παρίσι. Και παρόλο που δεν ξέρουμε πώς έφτασαν τα όπλα αυτά στο Παρίσι, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέσουμε και να παλύψουμε τα πλεονάσματα. Και μάλιστα οι πρόσφατες επιθέσεις στο Παρίσι δείχνουν πόσο σημαντική είναι η σωστή διαχείριση των όπλων και πυρομαχικών παντού, γιατί κυκλοφορούν παράνομα ακόμη πολλά όπλα στη Βοσνία Ζεγοβίνη και οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν την ευθύνη για 17 αποθήκες πυρομαχικών και 13 αποθήκες ε, όπλων που βρίσκονται ε, ανά την πόλη, ε, ανά την χώρα. Και μάλιστα ένα μεγάλο τμήμα του είναι για τη χρήση του στρατού τη Βοσνίας Ερζεγοβίνη. Τα περισσότερα όμω περιμαχικά και όπλα είναι παροχημένα, είναι πλεονασματικά και θα πρέπει να παραπληστούν και να χρηστευτούν. Και μάλιστα η διεθνή κοινότητα προσπαθεί να πείσει τους, τις ένοπλες δυνάμεις της Βοσνίας Ερδεγοβίνης να χρηστεύσουν τους σωρούς αυτούς των αποθεμάτων και να αυξηθεί ο βαθμός της ε, διαχείρισης, της διάθεσής τους. Συνεχίζουμε λοιπόν ε, την προσπάθεια της αύξησης της ασφάλειας, κυρίως των ε, στρατιωτών που χειρίζονται την ασφάλεια αυτών των χώρων και σίγουρα θα πρέπει να αποτρέψουμε τα πυρομαχικά και όπλα αυτά να φτάσουν σε λάθος χέρια και να τροφοδοτήσουν ε, η τρομοκρατία και βία είτε στη Βοσνία Ζεγοβίνη είτε παντού. Και μετά το καλοκαίρι θα ξαναξεκινήσουμε την ετήσια συζήτηση για την πιθανή ε, παράταση της εκτελεστικής εντολής της επιχείρησης Αλτέα. Και χρήσιμο θα ήταν γιατί εξακολουθούμε ε, να έχουμε μικρές αλλά πραγματικές δυνατότητες για επαναφορά της αθωνατικής βίας. Γι' αυτό θα πρέπει η ΑΛΤΕ να συνεχιστεί προκειμένου να αποφευθεί η διολύστηση προς μια χαοτική κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έτοιμα να επέμβει σωστά, κατάλληλα και σχετικά σύντομα και να αναπτύξει εφέδρους και ενισχύσεις προκειμένου να έχει διάφορες επιχειρήσεις για να εξασφαλίσει ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Για παράδειγμα, ε, προστασία αεροδρόμων, διαχείριση αποθηκών, πυρομαχικών και ακριβικών και κυρίως ε, διαχωρισμό πλήθους ε, βίαιου σε πόλεις με παρουσία διαφορετικών αθλητικών κοινοτήτων. Ε, παραλαμβάνω, οι πολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις προσπάθειές μας για εκπαίδευση και δημιουργία ικανοτήτων. Βέβαια, οι ένοπλε δυνάμει τη Βοσνία Ερζεγοβίνη επαναλαμβάνουν από του ε, καλύτερου ε, και πιο ε, οργανωμένου κλάδου και θεσμού τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και πραγματικά είναι το καμάρι του έθνου. Βέβαια, υπάρχει κάποιο κίνδυνο αστάθεια ακόμη στη χώρα αυτή. Και ακριβώ εξαιτία αυτή τη αστάθεια υπάρχει πάντα πιθανότητα έξαρση τη βία. Και βέβαια ο κίνδυνος για επέκταση αυτή στη χώρα είναι μικρός, αλλά οι συνέπειες ε, μιας τέτοιας κατάστασης ε, θα ήταν πολύ σοβαρές. Γι' αυτό η παρουσία μιας ε, ευρωπαϊκής δύναμης με εκτελεστική εντολή είναι επιθυμητή, όχι μόνο για να αποτρέψει το ξέσπασμα βίας στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, αλλά και κυρίως να αποτελέσει πηγή εμπιστοσύνη σε ένα πληθυσμό που έχει πολλές μνήμες από πολύ επώδυνες συγκρούσεις του παρελθόντος. Αυτά σας ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στρατμό. Μπράτσο, στρατηγέ μου. Κύριος Γκάλλος, παρακαλώ, για να αρχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά. Γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ, για την παρουσίαση και τα καθήκοντα που αναλαμβάνετε. Capacity Building and Training το ονομάσατε. Το σύνολο των καθηκόντων σας, ανάπτυξη δυνατοτήτων και κατάρτιση. Πρόκειται νομίζω για μια συμβολή στην ενσωμάτωση που μπορούμε να προσφέρουμε στο πλαίσιο του στρατού. Η σύνθεση των σωμάτων που λέτε ότι έχετε εκεί, τρία σώματα ισοδυναμεί λίγο πολύ στην τάξη μεγέθους των τριών ε, εθνοτικών ομάδων ή είναι πιο μεγάλη Φερρυπίνη, η Βοσνιακή ομάδα, οι Σέρβοι λιγότεροι ή οι Κροάτες. Μπορείτε να μας πείτε λίγο για τη σύνθεση. Και θα ήθελα να ρωτήσω πώς αξιολογείται την κατάσταση. Υπάρχει στην αλυσίδα διοίκησης αξιοπιστία υπάρχει η έννοια της αφοσίωσης και πίστης. Διαπιστώνεται κάτι τέτοιο ή υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένω. Εάν προκύψει κρίση. Ή αν σε ένα από τα κρατήδια όπως τη Ρεπουμπλίκα Σέρψκα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε το ενδεχόμενο να προκύψουν δυνάμεις ασφαλής της ε, Ρεπούμπλικα Σερψκά, τις οποίες θα μπορούσε να ακολουθήσει αυτό το σερβικό κομμάτι του στρατού της Βοσνίας. Βλέπετε λοιπόν κάποιο τέτοιο κίνδυνο ή νομίζετε ότι η ενοποίηση είναι τόσο ισχυρή που να επιτρέπει και την υπερπίδηση των πολιτικών κρίσεων. Και θεωρείτε ότι η παρουσία σας με τις δυνάμεις που έχετε είναι επαρκή. χρειάζεται ενίσχυση, χρειάζεται ενδεχομένω να περιοριστεί. Πώ το αξιολογείτε. Ευχαριστώ. Φρόιντ. Ευχαριστώ. Είμαι Αυστριακό. Χώρα, από χώρα η οποία επίση έχει συμβάλει πολύ στη Βοσνία για μεγάλο διάστημα. εφόσον επικεντρωθήκατε κυρίως στις στρατικές πτυχές της κατάστασης στη Βοσνία. Εγώ θα ήθελα. Περιμένω να ακούσετε. Θα ήθελα να ρωτήσω μια περισσότερο πολιτική ερώτηση εγώ. Τα κυριότερα προβλήματα στη Βοσνία που τα επικεντρώνεται, πού θα επισημαίνεται. Από το 95 αν δεν απατώμε με τη συνθήκη των Παρισίων, ή κάποια χρόνια μετά, 98, το 95, πότε ήταν. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, περίπου 20 χρόνια πέρασαν από τότε πάντως. Ξέρετε, μεταξύ Είχαμε τρεις, είπα τους εκπροσώπους αυστριακούς που παρακολουθούσαν την κατάσταση. Από αυτούς λοιπόν ενημερώνομαι ότι ήταν τόσο περιορισμένη η πρόοδος στο πολιτικό πεδίο με τα φαινόμενα της διαφθοράς και τα άλλα. Και γι' αυτό σας ερωτώ, εάν έχετε κάτι εσείς να απαντήσετε σε αυτό και ότι είστε βέβαια στρατιωτικός διοικητής, έχετε ζήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στη χώρα και ίσως μπορείτε να αξιολογήσετε την κατάσταση πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρτεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Στρατηγιά. Καλώς ήρθατε. Με βεβαίως πως ε, οι θεωρητικές δυνάμεις θα επιτελέσουν το έργο τους με το μέγιστο επαγγελματισμό οπουδήποτε ε, αποσταλούν και κυρίως να πρόκειται για Βρετανούς αξιωματικούς. Δεν θα προσπαθήσω να σας ε, προσελκύσω σε μια συζήτηση για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία όπως γνωρίζετε ε, εκβάθρον απορρίπτω. θεωρώ ότι και την προσοχή αλλά και τους πόρους μας παρεκτρέπει από το κύριο ζήτημα που είναι το ΝΑΤΟ είναι πολιτικό σχέδιο η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνα. ένα σχέδιο ενοποίηση το οποίο δεν υποστηρίζουμε πολλοί από εμά. και νομίζω ότι έχετε τον μη αξιόφθονο, το μη αξιόφθονο καθήκον να ε, μας πείθετε, να προσπαθείτε να μας πείθετε κάθε φορά χωρίς επιτυχία όμως. Βάση περιπτώσει υπάρχει ένα άλλο σοβαρό σχέδιο που με ενδιαφέρει και αφορά την βιωσιμότητα του κράτους της Βοσνίας και Ε, Μιλήσατε για την περίοδο μετά τον Τζέιτον και θα ήθελα σε αυτό ακριβώς να επικεντρωθούμε γιατί έχει περάσει πολύ καιρό όντω. Μια δύο ερωτήσει λοιπόν. Πού θα εντοπίσετε τον κύριο κίνδυνο για τη σταθερότητα του κράτους σε σχέση με την αποστολή που έχει αναπτυχθεί στη Βοσνία και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι υφίσταται πραγματικός κίνδυνος ή εκφράζουν πραγματικό κίνδυνο οι όμοροι, τα όμορα κράτη της περιοχής. Επίσης, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα της αποναρκοθέτησης. Η Βοσνία βεβαίως έχει διασπαρεί με ε, χερσαίες νάρκες. Πρέπει τώρα πια να αποδοθούν τα εδάφια αυτά καθαρά για χρήση, κατάσταση και χρήση και αξιοποίηση. Θεωρείτε λοιπόν ότι έχει όντως γίνει σωστά η αποναρκοθέτηση στην ε, Βοσνία και Ερσεγοβίνη. Και κάτι ακόμη στο οποίο δεν αναφερθήκατε τόσο διεξοδικά. Το ότι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φυτόριο τζιχαντιστών. Αν ανατρέξουμε στις αρχές αυτής της ε, αντιπαράθεσης, ήταν αρκετά σαφές ε, το φαινόμενο της διαστηριοποίησης τσιχαριστών στην περιοχή. Θέλω να δούμε τι είδους παρακαταθήκη έχουν αφήσει. Είναι μόνο ή και άλλα ζητήματα. Μπορείτε να αναφερθείτε πιο δεξιωτικά. Ευχαριστώ. Ράδος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε, κυρίες και κύριοι, στρατηγέ. Ένα από τα καθήκοντα της επιχείρησης Αλτέα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι η και αλλα ζητηματα μπορειτε να αναφερθειτε πιο δεξιδικα ευχαριστω ραδος ευχαριστω κυριε προεδρε κυριε κυριες και κυριοι στρατηγε ενα απο τα καθηκοντα της ε, γενικής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Η στρατηγική αποστολή δεν είναι ο καλύτερος τρόπος ε, να στηριχθεί η γενική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Και περίπου 20 χρόνια κρατάει αυτό το τμήμα της αποστολής, ε, αν συμπεριλάβουμε και την εποχή που είχαμε την νατοϊκή αποστολή. Βέβαια φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι με τους οποίους στηρίζεται αυτή η επιχείρηση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα των ε, ριζοσπαστικών Ισλαμιστών στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και μάλιστα τα μηνύματα που ακούσαμε σε τζαμιά στη διάρκεια των ε, λειτουργιών ήταν πολύ ανησυχητικά. Και φαίνεται ότι υπάρχει ένας εκφοβισμός στη Βοσνία Ζεγοβίνη όλων όσων είναι κατά του ριζοσπαστικού Ισλάμ και φαίνεται ότι συνεχίζεται, η στρατολόγηση μαχητών για την αποστολή στη Συρία υπέρ του ε, Ισλαμικού κράτους. Και Ακόμη και στις ε, αρχές της Βοσνίας ε, Ζεγοβίνης υπάρχουν πολλοί που τάσσονται υπέρ του ριζοσπαστικού Ισλάμ και στηρίζουν ακόμη και την ε, τρομοκρατία που είναι ένα τμήμα των δραστηριοτήτων του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Και μάλιστα πολύ ανοιχτά και ηχηρά λένε ότι η Βοσνία με τις δυνάμεις της και την οργάνωση δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσει 3.000 ε, ε, δυνητικούς τρομοκράτες που με βάση τις δηλώσεις της ίδιας της Βοσνίας ήδη έχουν βρεθεί σε διάφορα πεδία μάχης στη Συρία και μάλιστα μερικοί έχουν και επιστρέψει από τη Συρία. Ερωτώ λοιπόν σε ποιο βαθμό η Eurofor ε, Altea και η επιχείρησή σας ασχολείται με το πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Λούζιν. Σας ευχαριστώ. Μιλήσατε για την ε, ανήσυχη κατάσταση που επικρατεί και μιλήσατε, αν κατάλαβα σωστά, και για κοινωνικές ε, ανησυχίες, αναταραχές. Και συζητήθηκε αυτό ιδιαίτερος, καθώς και τα συμπεράσματα, η σύγκριση με τα περιστατικά το Παρίσι, όλα κινήθηκαν πολύ γρήγορα προς μια κατεύθυνση και κατέληξαν στο συμπέρασμα μιας μεγάλης φασιστικής πρόκλησης. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στα αίτια των ανησυχιών αυτών. Είπατε ότι οι αιτίε δεν έχουν αξιολογηθεί και δεν έχουν τροποποιηθεί. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να συζητήσουμε ποια είναι τα αίτια αυτών των περιστατικών είτε πρόκειται για διαμαρτυρίες ε, του κόσμου, είτε για νόμιμες διαμαρτυρίες ενδεχομένω του κόσμου. Εγώ πάντα αυτό που υποστηρίζω είναι το εξή. Στο... Στις ε, διαμαρτυρίες, όταν υπάρχει βία, αυτό είναι θέμα της αστυνομία. Εδώ η όλη η συζήτηση εστιάζεται σε μια στρατιωτική πρόκληση. Ερωτώ λοιπόν, τα καθήκοντα του στρατού εκεί πώς πρόκειται να οριστούν στο μέλλον. Διάβασα κάπου ότι όταν ήταν πολύ οξύες αυτές οι διαμαρτυρίες, ο ε, ε, πρεσβευτής ε, του ΟΗΕ στη Βοσνία κάλεσε κατά των περιστατικών αυτών, κατά των διαμαρτυριών. θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και αυτό ως λύση στις τρέχουσες ε, καταστάσεις. Και τι δυνατότητες ε, έχουμε στην προκειμένη περίπτωση. Τι σκέφτεστε. Σας ευχαριστώ. Λέει Πρόεδρος, θέλει κανείς να μιλήσει εξ ονόματα των πολιτικών ομάδων. Αν όχι, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον στρατηγό Μπράτσο τώρα για να απαντήσει στο πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Έχετε το λόγο. Κυρίε και κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ερωτήσει σα. Καταρχά, προ τον κύριο Γκάλερ και τα ερωτήματά μου για τη σύνθεση των ένοπλων δυνάμεων τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Οι ένοπλε δυνάμει είναι λίγο πολύ κατά αναλογία του πληθυσμού, τη σύνθεση του πληθυσμού, παρά το γεγονός ότι η πρόσληψη των αξιωματικών τώρα γίνεται με μη εθνοτικά κριτήρια. Μη. Δηλαδή βασιζόμαστε σε αξιοκρατικά κριτήρια, αποκλειστικά πλέον. Αυτό είναι πάρα πολύ τολμηρό βήμα αλλά αληθεύει. Στις ένοπλες δυνάμεις όντως υπάρχουν ακόμα ε, μονάδες που βασίζονται ε, στην εθνοτική σύνθεση της εκάστοτε περιφέρειας και περιοχής. Ρωτήσατε για την αξιοπιστία της αλυσίδας ε, εντολών. Και θέσατε ερωτηματικά σε ό,τι αφορά την δυνατότητα των εθνοτικών ομάδων να προσπίσουν το κοινό συμφέρον. Οι αξιωματικοί που έχω γνωρίσει στις αναπλές δυνάμεις της Βοσνίας πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ δεσμευμένοι για το σύνολο του στρατιωτικού σώματος και επιδεικνύουν ε, ιδιαίτερη περηφάνεια για την οργάνωση του σώματος. Είναι πάρα πολύ περήφανοι σε ό,τι αφορά αυτά που συμβάλλουν και συνεισφέρουν στο διεθνές προσκήνιο. Και αυτό τους δίνει μεγάλη αξιοπιστία ως αθλητικούς. Θα έλεγα ότι υπάρχουν σχετικά σταθερές λοιπόν συνθήκες. Είναι απόλυτα αξιόπιστοι σε τέτοιες συνθήκες σταθερότητας. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε σε ποια φάση θα μπορούσε να διαλυθεί αυτή η σταθερότητα, αυτή η κατάσταση. Αλλά θεωρώ ότι σε περίπτωση που αν ε, υπήρχε κάποια εθνοτική τριβή στο μέλλον, το οποίο το πευχόμαστε, υποπτεύομαι ότι οι πιέσει ε, για τους στι στις δυνάμει θα ήταν κάποια στιγμή υπερβολικά μεγάλες και θα έπρεπε να καταφύγουν στην προάσπιση των δικών τους ανθρώπων. Αλλά στην παρούσα φάση οι ένοπλες δυνάμεις στη Βοσνία Ζεγοβίνη επιδεικνύουν ιδιαίτερη αλληλεγγύη και επαγγελματικά προσόντα. Για τον κύριο Φρόιντ, επιστήσατε την προσοχή μας ε, στο... στη μεγάλη χρονική περίοδο για την οποία βρισκόμαστε εκεί και στη μεγάλη περίοδο σταθεροποίησης και στην επίμονη φύση κάποιων ιδιαίτερων δυσκολιών που χαρακτηρίζουν την Βοσνία ζεβοβινη Οι πιο πολλές εκ των οποίων ασφαλώς πηγάζουν από την εθνοτική φύση της σύνθεσης της χώρας. Θα συμφωνούσα μαζί σας λοιπόν. Και νομίζω ότι αυτό μοιραία μας οδηγεί στο επόμενο ερώτημα. Κατά πόσον είναι απαραίτητο να υπάρχει στρατογική υπομονή στο σημείο αυτό. Προφανώς παίρνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η σταθεροποίηση της κατάστασης. Βλέπουμε κάποιες μικρές ενδείξεις πολιτικής οριμότητας, όπως ανέφερα, κάποιες ενδείξεις που δικαιολογούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που περιμέναμε δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και θα είναι δύσκολο να επιτευχθούν σε μια χώρα που μαστίστηκε από μια τέτοια διαμάχη σύγκρουση όπως η Βοσνία Ζεγοβένη παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Είναι θέμα αλλαγής γενιάς ουσιαστικά το να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Δουλεύουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά καλό θα ήταν να ακολουθηθεί η αρχή της πρόληψης σε ό,τι αφορά τις ε, διαταξίες ασφαλείας. Και φυσικά οι ένοπλες δυνάμεις της Βοσνής Ερζεγοβίνης δεν διαδραματίζουν ρόλο στην εσωτερική σταθερότητα. Στην εσωτερική σταθερότητα. Οι μοναδικές λοιπόν στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες είναι ικανές να διαδραματίσουν τον συγκεκριμένο ρόλο, είναι οι δυνάμεις της UFOR. Δεν ξέρω αν απαντάω έτσι απόλυτα στο ερώτημά σας, αλλά αυτό που λέω είναι ότι η ισορροπία όσο έχει σήμερα ενδεχομένως να μην σημειώνει ιδιαίτερη πρόοδο, όχι ιδιαίτερα ε, γρήγορα, αλλά τουλάχιστον είναι αρκετά σταθερή ως ισορροπία. Καλό θα ήταν να μην διταραχθεί. Για τον κύριο Φανόρτεν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, εμπιστοσύνη που εκφράζεται στην Βρετανική ηγεσία, στρατηγική ηγεσία. Μιλήσατε για την βιωσιμότητα του κράτους της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και ασφαλώς αυτό αποτελεί ένα απόλυτα πολιτικό ζήτημα. Όντως, υπάρχουν πιέσεις στο ιστορικό του κράτους και υπάρχουν κάποιες δυνάμεις οι οποίες ενδεχομένως να διαλύσουν αυτή την σταθερότητα και την ισορροπία. Πρόκειται για μια πολιτική παρατήρηση, δεν είναι δικό μου, δική μου αλλά πιστεύω ότι η εστίαση στην ε, ένταξη στην Ευρώπη για την οποία συζητάνε όλοι οι πολιτικοί από όλες τις εθνικές ομάδες αποτελεί μια στατική πολιτική ένταξη. Ένα στατικό πολιτικό φαινόμενο το οποίο αποτελεί και κινητήριο δύναμη για την περαιτέρω συνοχή της χώρας. Και θεωρώ λοιπόν ότι είναι θετική η εξέλιξη αυτή. Αναμφίβολα υπάρχουν ιστορικές πιέσεις στη χώρα, καθώς η χώρα κινούνται προς την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Νομίζω ότι στην πορεία λοιπόν αυτή προς την Ευρώπη υπάρχει περιθώριο μείωσης και αποσυμπίεσης των τάσεων και των μετάσεων αυτών για την... προκειμένου να ξεπεραστούν οι τριβές. Όπως σας είπα, ένα σταθερό, μια σταθερή ισορροπία, η οποία ενδεχομένω να μην κινείται αρκετά γρήγορα, αλλά είναι αρκετά σταθερή, είναι προτιμητέα από μια κατάρρευση τη σταθερότητα αυτή. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να ξεσπάσει εθνική, εθνική βία. Το Φεβρουάριο λοιπόν είδαμε μια τέτοια πιθανότητα να διαγράφεται, όπου ουσιαστικά κοινωνικά ζητήματα, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα διατάραξαν την κατάσταση και χρησιμοποιήθηκαν από άτομα τα οποία προωθούσαν την εθνοτική τους, εσωτερική πολιτική τους ατζέντα. Αυτό φυσικά υπονομεύει τη σταθερότητα και φυσικά ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα είναι να στοχευτεί ο πυρήνας του προβλήματος οι κοινωνικές, ε, οικονομικές αιτίες. Αυτό ασφαλώς αποτελεί έργο της κυβέρνησης. Αλλά όπου υπάρχει πιθανότητα ξέσπασμα εκνοτικής βίας, θεωρώ ότι καλό είναι και σόφρον είναι να υπάρχουν κάποια περιορισμένα μέτρα προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα αντίδρασης, προκειμένου να μην ε, πάρει υπερβολικές διαστάσεις αυτή η βία. Ρωτήσατε ποιες είναι οι απειλέ από τι γειτονικέ χώρε. Στην παρούσα φάση αυτό δεν φαίνεται να αποτελεί ένα στοιχείο, ένα παράγοντα στην ασφάλεια τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Από ό,τι φαίνεται, οι γειτονικέ χώρε υποστηρίζουν την αρχή τη σταθερότητα στο εσωτερικό τη χώρα αυτή. Επίση, ε, ρωτήσατε για θέματα Ισλαμικού εξτρεμισμού. Αληθεύει ότι ε, διάφορα άτομα έφυγαν από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη ως ε, μαχητές και πήγαν στην Συρία, στο Ιράκ για να πολεμήσουν. Και φυσικά ο κόσμο ανησυχεί τι θα γίνει όταν θα επιστρέψουν ενδεχομένω αυτά τα άτομα στην Βοσνία Ζεγοβίνη. Αυτό ισχύει και για όλη την Ευρώπη άλλωστε. Είναι ένα αληθινό ενδεχόμενο. Οι εκτρεμιστέ να αποτελέσουν παράγοντα για διεθνικές ε, εντάσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν οι ε, υπηρεσίε, οι ε, μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας στην Σερβία να παρακολουθούν το φαινόμενο αυτό επισταμένως. Νομίζω ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ενότητα μεταξύ των αισθηματικών ομάδων αναφορικά με την ανάγκη να συλληφθούν τέτοιοι εξτρεμιστές Ισλαμιστές. Για να απαντήσω στον κύριο Ράπτος τώρα. Η στρατιωτική αποστηλή, είπατε, δεν αποτελεί τον καλύτερο τρόπο υποστήριξη τη γενικότερη στρατηγική την οποία έχουμε για τη Βοσνία Ζεγοβίνη. Υποδείξατε δε το φαινόμενο του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Στρατιωτική Αποστολή δεν ε, μειώνει σε καμία περίπτωση του στρατηγικούς μας στόχους και ακόμα και μια περιορισμένη ε, ικανότητα και αν έχει να αποτρέψει ένα ξέσπασμα εθνοτικής βίας, θεωρώ ότι αποτελεί κάτι στατικό. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την ε, τοποθέτησή σας. Η παρουσία ριζοσπαστικών ισλαμικών στοιχείων εντός του πληθυσμού αποτελεί πηγή ανησυχία. Και όπως έχουμε ήδη συζητήσει, αυτό είναι κάτι που του παρακολουθούν οι υπηρεσίες ασφαλείας της Βοσνίας Αρζεγοβένης. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν εναπόκειται στις ε, αρμοδιότητες ε, των υπηρεσιών ασφαλείας της ε, Βοσνίας Ερζεγοβίνης, σε περίπτωση δηλαδή που υπάρχει παράνομη δραστηριότητα. Για την κυρία Λόζεν, σας ευχαριστώ και εσάς για τα ερωτήματα που μου θέσατε. Είπατε ότι συγκρίνω τις κοινωνικές αναταραχές στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με το Παρίσι. Δεν ήταν αυτή η σύγκριση. Εγώ απλά ανέφερα ότι κάποια από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιήθηκαν στις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι είχαν προέλθει από το, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Το πώς μεταφέρθηκαν είναι εντελώς αβέβαιο. Αλλά αυτό που ήθελα να θίξω είναι το εξής, ότι δεν υπάρχουν πολλά εκρηκτικά στη Βοσνία Ζεγοβίνη που δεν χρειάζονται για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και που δεν προστατεύονται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις είναι κάτι το αρνητικό και θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό λοιπόν εξετάζουμε. Οι 17 αποθήκες εκρηκτικών ε, εξετάζονται προκειμένου με πιο σωστό τρόπο να δημιουργηθούν, να επισκευαστούν κτίρια προκειμένου να είναι πιο ασφαλή τα εκρηκτικά. Και φυσικά φροντίζοντας να αποθηκεύονται τα εκρηκτικά σε λιγότερες εγκαταστάσεις, μπορούμε να μειώσουμε και τα ρυθμό των στρατιωτών που τα προστατεύουν και τα φυλάνε. Το οποίο ταιριάζει φυσικά με τους γενικότερους στόχους μας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του δυναμικού. Μιλήσατε τώρα για την αξιολόγηση των προβλημάτων που προκαλούν τις αναταραχές, που προκάλεσαν τις αναταραχές του προ, τον προηγούμενο Φλεβάρι. Οι δείκτες ε, καταδεικνύουν ότι τα αίτια είχαν να κάνουν με κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ανεργία, κοινωνική, κοινωνικές συνθήκες. Υπάρχει μια κάποια απογοήτευση σε ό,τι αφορά την ε, έλλειπη εξέλιξη και πρόοδο αναφορικά με τα ζητήματα αυτά. Άρα ο κόσμος έχει κάποιο δίκιο, αλλά φυσικά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του να διαδηλώνει κανείς ειρηνικά για να, προσ... να προασπίζει τα πολύ σεμιτά στοιχεία αυτά και την βία που ξέσπασε και η οποία ασφαλώς εκμεταλλεύτηκε μετά αποτέλεσε αντικείμενο εκμετάλλευσης από άλλους που είχαν άλλα κατά νου και δικά τους προσωπικά συμφέροντα. Νομίζω ότι απάντησα έτσι στις περισσότερες ερωτήσεις που μου τέθησαν και ευχαριστώ να επανέλθω. Σας ευχαριστούμε στρατηγέ. Περάμε τώρα στο δεύτερο γύρο της συζήτησης. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πράδρα, Έχω δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ε, πρώτοι αναφέρθηκαν και συνάδελφοι και εσείς στρατηγέ. Σε περίπτωση κλιμάκωσης της κατάστασης, δηλαδή ξεσπάσματος βίας, η έξαρση των ε, ταραχώρων όπως είχαμε πέρυσι το Φεβρουάριο, δεν κάνω λάθος, και σε περίπτωση αποτυχίας των βοσνιακών αρχών να ελέγξουν την κατάσταση. Έχουμε εμείς ε, δυνατότητες, ικανότητες αντίδρασης. Δηλαδή θα μπορέσετε να αναπτύξετε αμέσως και επιτόπου για μια συντονισμένη δράση κάποιες ε, στρατιωτικές μονάδες. Δεύτερο, ε, με ενδιαφέρον παρατηρήσαμε ότι οι Ρώσοι απήχαν ε, στο θέμα, στη συζήτηση τον Νοέμβριο για την παράταση της εντολής U4. Δεδομένης παρούσας κατάσταση των σχέσεων ευρωπαικη Ευρωπαϊκή Ένωση-Ρωσία. Μήπω φέτο πιστεύετε ότι η Ρωσία θα υποβάλει και βέτο στην παράταση τη εντολή. Κάτι που θα οδηγήσει σε τερματισμό τη επιχείρηση Αλτέα. Οπότε ουσιαστικά οι Ρώσοι θα ε, αποπέμψουν την, ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση από την επικράτεια της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Ξέρω δεν είστε πολιτικός, αλλά θα ήθελα να σχολιάσετε τη πιθανή αυτή κατάσταση και τις συνέπειες που θα έχει επιτόπου. Μπορούμε να υπολογίσουμε σε οποιαδήποτε συνεργασία με τη Ρωσία στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ. Αν δεν θέλει άλλος κανείς το λόγο, θα ήθελα και εγώ να θέσω κάποιες ερωτήσεις στρατηγέ. Η επιχείρηση U4 Altea είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα των ε, δεσμών ε, των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με τις ε, επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Χρησιμοποιώντας το μηχανισμό Βερολίνο ΣΥΝ. Μπορείτε να μας ε, πείτε δύο λόγια για αυτές τις συνέργειες ανατοικών και ενωσιακών επιχειρήσεων, γιατί έχουμε πολλούς νέους ευρωβουλευτές και ίσως δεν γνωρίζουν αυτές τις διασυνδέσεις. Δεύτερον, πιστεύετε ότι υπάρχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ της ε, ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με την κατάσταση στη Βοσνία και την Ερζεγοβίνη. Δηλαδή, ε, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε επιπλέον ταραχές ε, στην Σερβική Δημοκρατία, στη Ρεπούμπλικα Σέρψκα ή δημιουργήθηκαν φαινόμενα συναφή με αυτό που συνέβη στην Ουκρανία. Επίσης, ε, είπατε ότι πολεμοφόδια και πυρομαχικά από τη Βοσνία φαίνεται ότι κατέληξαν στο Παρίσι και χρησιμοποιήθηκαν εν μέρη και στις επιθέσεις του Παρισιού. Κάποια μέσα μαζικής ενημέρωση έδωσαν άλλα στοιχεία ότι από την Τσετσενία προήλθαν αυτά τα πολεμοφόδια και πυρομαχικά. Γνωρίζουμε ότι για πολλά χρόνια η Βοσνία ήταν ε, εστία πολλών ριζοσπαστών, Ισλαμιστών και Μοχαβητών. Και ξέρουμε και σήμερα ότι πολλοί νέοι της Βοσνίας στρατολογούνται από το Ισλαμικό κράτος και πηγαίνουν να αγωνιστούν στο πλευρό του Ισίλ. Πώς πιστεύετε ότι η δική σας επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, κύριε Κούκαν, αν έχουμε τις ικανότητες αντίδραση σε περίπτωση έξαρσης της βίας στη Βοσνία Ζεγοβίνη. Μόνο 600 στρατιώτες ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ε, και οι δυνατότητες μας για άμεση αντίδραση είναι περιορισμένοι. Μάλιστα τον περισμένο Φεβρουάριο είχαμε τέτοιες ταραχές και ίσως ε, έτσι μπορούμε να δούμε με βάση τη συνέβη πέρυσι πόσο άμεσα μπορούμε να αντιδράσουμε. Στο Μοστάρ είχαμε κάποιες, είδαμε κάποιες ομάδες διαδηλωτών που διαδήλωναν ε, και στις δύο πλευρές της ε, οροθετικής γραμμής, της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ των δύο εθνοτήτων ε, στην πόλη του Μοστάρ. Και οι διαδηλώσεις άρχισαν να παίρνουν ένα πιο δύο χαρακτήρα. Ο διοικητής ξεκίνησε ε, κάποιες ε, ενέργειες και είπε να αναπτύξει ένα τμήμα της στρατιωτών της Αλτέα ανάμεσα στις δύο εθνοτικές μονάδες ώστε να τους κρατήσει ε, σε απόσταση προκειμένου να κατευναστούν τα πνεύματα και να επικρατήσουν οι πιο ψύχρεμοι και όχι θερμόεμοι. Και νομίζω ότι αυτή ήταν πολύ λογική και κατάλληλη, κατάλληλη ενέργεια για να δώσουμε κάποια, ε, κάποιο περιεχόμενο σε αυτή την εκτελεστική εντολή. μάλιστα έχουμε και σε επιφυλακή τρία εφεδρικά αποσπάσματα που μπορούν σε, να αναπτυχθούν σε περισσότερα από μία περιοχές. Πάντως, αν γενικευτούν οι προοπτικές ε, για ξεσπάσματα βίας και έντονες διαδηλώσεις, θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε κάποιες βασικούς ε, οδικούς άξονες ή αεροδρόμια με τη διεθνή παρουσία. Και έχουμε στην επιχείρηση Αλτέα διάφορα σχέδια εκτάκτου ανάγκης για τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε επίσης και ένα τάγμα επιχειρησιακών εφεδριών για ευρύτερες ε, ενέργειες. Πάντως ε, το επιχειρησιακό μας σχέδιο προβλέπει και πρόσβαση και σε τρία εφεδρικά τάγματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα όμως τάγμα ε, σε τέτοιες επιχειρήσεις. Οπότε δεν υπάρχουν αρκετές εφεδρίες και αν εμπλακούμε σοβαρά στην εξασφάλιση προστασίας και ασφάλειας σε διάφορες ζώνες, ιδιαίτερα ε, κοντά σε αποθήκες ε, με πυρομαχικά και πολεμοφόδια, πολύ γρήγορα θα εξαντληθεί το δυναμικό μας και η ικανότητα αντίδρασης. Και θα πρέπει στην Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας να εξεταστεί η πιθανότητα χρήσης ε, ευρωπαϊκών ομάδων μαχητικών στην Αλτέα. Τώρα, μήπως η προηγούμενη εποχή των Ρώσων είναι πρελούδιο σε ένα μεταγενέστερο βέτο εξαιτία τη ε, όξυνση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα είναι αν ε, αποχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σταθεροποιητικό αντίκτυπο στη Βοσνία, μια τέτοια αποχώρηση θα αποβεί προς όφελος της Ρωσίας. Οπότε αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Τώρα, ε, σε, στην περίπτωση αυτή συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία και έτσι πρέπει να γίνεται. Σε περίπτωση όμως που έχουμε κάποια στοιχεία ριζοσπαστικού Ισλάμ στη Βοσνία Ζεγοβίνη, αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο και ενδιαφέρει και τη Ρωσία και πολλά άλλα έθνη. Οπότε, το να παρακινούμε να δημιουργούμε πρόσφορα έδαφος για αστάθεια και ανασφάλεια, ε, κάτι που θα τροφοδοτήσει ουσιαστικά τέτοια εξτρεμιστικά και ριζοσπαστικά φαινόμενα, αυτό δεν είναι ούτε προ όφελο τη Ρωσία ούτε κανένα άλλο κράτο. Οπότε είναι προ αβεβαίω συμφέρον η καλύτερη συνεργασία με τη Ρωσία γιατί, για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια απειλή που μπορεί να στραφεί απέναντι σε όλε τι κοινωνίε. Επίσης, κυρία Πρόεδρε, μιλήστε για τις διασυνδέσεις των ατοικών επιχειρήσεων με τι ευρωπαϊκές. Είναι ένα παράδειγμα ε, ε, των συμφωνιών που στηρίζονται στο μηχανισμό Βερολίνο ΣΥΝ. Η Αλτία είναι τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγαστής συνεργασίας του ΝΑΤΟ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα φαίνεται ότι είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματική αυτή η χρήση του προσωπικού και των πόρων διοίκησης. Και σε μια εποχή που το ΝΑΤΟ επικεντρώνεται σε θέματα περισσότερο συλλογικής άμυνας, άρθρου 5, το μείζον θέμα του συντονισμού των στρατηγικών προσπαθειών στα πλαίσια του άρθρου 5 της συλλογική άμυνας ε, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο, μεγαλύτερες ευκαιρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει περισσότερες επιχειρήσεις σταθεροποίηση. Και είναι κρίμα που οι συμφωνίες Βερολίνο-ΣΥΝ δεν μπορούν να παραταθούν και για πολιτικούς λόγους και σε άλλες περιοχές. Πάντως, θα πρέπει να προσέξουμε και να αποφύγουμε επικαλύψεις των προσπαθειών μας με τον ΝΑΤΟ. Γιατί το ΝΑΤΟ σίγουρα είναι μια οργάνωση που ασχολείται με συλλογική άμυνα μεγάλης εμβέλειας και μεγάλης εμβέλειας επιχειρήσεις σταθεροποίησης, όπως το Αφγανιστάν. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται με μικρής εμβέλειας σταθεροποιητικές επιχειρήσεις, όπως είναι η Αλτέα, για παράδειγμα. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ αποτελεσματική κατανομή και επιμερισμός ευθυνών. Ε, το ΝΑΤΟ ε, υιοθετεί μια πιο γενική ε, έποψη, αλλά πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι οργάνωση που θα προβλέπει τις βασικές προδιαγραφές εκπαίδευσης και τις προδιαγραφές για τις διάφορες επιχειρήσεις των κρατών μελών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις των προσπαθειών μας. Και φαίνεται ότι η χρήση των διαδικασιών του ΝΑΤΟ θα ήταν αποτελεσματικός τρόπος ε, για τις δραστηριότητες και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί να προβαίνει σε δικό της προσδιορισμό των αρχών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική με τη Ρωσία, πιστεύω ότι και εδώ θα πρέπει να εξασφαλιστεί στενή συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η ρωσική στρατηγική στην Ουκρανία είναι μια πιο σφαιρική στρατηγική και απαρτίζεται από πολλά στοιχεία ε, πολιτικής εξουσίας και όχι μόνο στρατητικής. Ενώ το ΝΑΤΟ είναι μια στρατητική οργάνωση. Οπότε, σε ό,τι αφορά την παροχή αρρωγής ε, στα μέλη του, προκειμένου να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αυτή την πιθανή ρωσική προσέγγιση. Εκεί θα μπορούσαμε να συμβάλλουμε σε στρατιωτικό επίπεδο, με συμβατικό και μη συμβατικό τρόπο, αλλά είναι περιορισμένες ε, οι δυνατότητές μας ε, για να βοηθήσουμε τα κράτη να προετοιμαστούν για τις άλλες πτυχές μια σφαιρική παραλαμβάνω στρατηγικής που έχει και πολιτικά ε, σκέλη και κοινωνικά. Εκεί πιστεύω ότι μπορεί να συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό ε, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά. Ρωτήσατε επίσης ε, κατά πόσο διαπιστώσαμε επιπλέον ταραχές ε, στην Ρεπούμπλικα Σέρψκα, στη Σερβική Δημοκρατία, μετά τα, τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Όχι, δεν διαπιστώσαμε τέτοιες ταραχές. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι εκεί η συμπεριφορά της Σερβίας. Και η Σερβία εστιάζεται στην ε, ένταξη της ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ θετικό και για την περιοχή. Δεν παίζει το ρωσικό χαρτί παρά τις ε, συνεχείς προσπάθειες της Ρωσίας να διευρύνει την ε, επιρροή της και προς τη χώρα αυτή. Πάντως είναι θετική η στάση της Σερβίας. Και συμφωνώ ότι η συνέχιση της ενταξιακής διαδικασίας ε, και της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων είναι πολύ θετική. Μιλήσατε για τους διαδρόμους ή τις διαδρομές που ακολούθησαν τα πυρομαχικά, τα πολεμοφόδια για να φτάσω στο Παρίσι μιλήσατε για το τσετσενικό διάβλο. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία. Ξέρω ότι μερικά πολεμοφόδια, μερικά πορομαχικά έφτασαν στο Παρίσι από τη Βοσνία. Τώρα με ποιο δρόμο έφτασαν. Αν πέρασαν και από τη Τσετσενία ή από άλλες περιοχές ε, δεν το γνωρίζω ούτε μπορώ να το σχολιάσω. Πάντως είναι ένα επιχείρημα επιπλέον που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης αντιμετώπισης ε, του θέματος των πλεονασματικών πυρομαχικών στη Βοσνία. Κύριε Βανόρντεν, αν δεν κάνω λάθος, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει φυσικά μια διαρκής ε, επιθυμία σε κάποια μέρη για να υπάρχει ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά και την ε, πολιτική ανασφάλεια. Μήπως αυτό ε, σχετίζεται με, το γεγονός αυτό. Δεν εξετάζεται ίσως επαρκώς. Θα ήθελα να τονίσω ένα στοιχείο το οποίο αναφέρατε για την έλλειψη αποθεμάτων για την έλλειψη ικανοτήτων ανταπόκριση σε περίπτωση ξεσπάσματος κρίσης. Και, την, ε, και σε περίπτωση που χρησιμοποιούνταν ένοπλες δυνάμεις. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχει παρουσία του ΝΑΤΟ στην Βοσνία και αν τα πράγματα πραγματικά σφίξουν, το πιο προφανώς θα ήταν να στραφούμε στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ. Εν συντομία, σε σχέση με αυτά που ρώτησε και ο κύριο Φανόρντεν και ήταν και στις πρώτες μου ερωτήσει. σύμφωνα με τι δικέ σα εκτιμήσεις στην ηγεσία της αποστολής αυτής, πιστεύετε ότι το μέγεθο είναι αρκετά, αρκετό της αποστολή για να ανταποκριθούμε σε περίπτωση ανάγκη ή χρειάζεται να υπάρξουν άλλες ε, απαιτήσει. Ευχαριστώ. Στρατηγέ, αν θέλετε να απαντήσετε για να κλείσουμε μετά. Σα ευχαριστώ πολύ. Για τον κύριο Βανόρντεν. Τα σχόλια μου για το δυναμικό μια μεγαλύτερη συνεργασία, στενότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ δεν στηρίζονται στην ιδέα του να αναζητούμε ρόλου για το ΝΑΤΟ για τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στρατιωτικές δομές, αλλά αναζήτηση της κατάλληλης, ε, του κατάλληλου επιμερισμού ευθυνών. Κατανομής αρμοδιοτήτων του ΣΥΠΗΝ, όπου υπάρχουν δυνατότητες βέβαια και στρατιωτικές δομές. Και όπως είπα, υπάρχει λογική να ρυθμίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πιο περιορισμένη συμβέλεια σε θέματα σταθεροποίησης μέσα στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της Ευρώπης, εκεί όπου είναι λιγότερο ισχυρά τα αμερικανικά συμφέροντα, τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αλλά αυτό με τη χρήση δυνάμεων εκπαιδευμένων σε επίπεδο ΝΑΤΟ, που μπορούν δηλαδή να τηρήσουν τις διαδικασίες αυτές. Αυτό νομίζω θα σήμαινε μια καλή κατανομή αρμοδιοτήτων και θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να λαμβάνει την ευθύνη για ευρύτερη, μεγαλύτερες επιχειρήσει εμβέλειας ε, επιχειρήσεις και δραστηριότητες. Τελευταία δεκαετία βεβαίω ιδιαίτερα επικεντρωθήκαμε σε μια πολύ απαιτητική επιχείρηση εκστρατεία στο Αφγανιστάν. Το γεγονό ότι μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει την ευθύνη για τις επιχειρήσει στη Βοσνία δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια τελείω ανεπιθύμητη εξέλιξη εν προκειμένου. Αλλά Πρέπει πιστεύω να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι περιττές δαπάνε στην ε, περίπτωση αυτή και άρα μία λογική ανάπτυξης αυτών των δομών ανεξαρτήτως της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν ε, περί τη δαπάνη, περί τη σπατάλη δυναμικού και πόρων εφόσον το ΝΑΤΟ μπορεί να τα κάνει εξίσου καλά. Μπορεί κανείς δηλαδή να πει ότι είναι πιο ε, αποτελεσματικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλεί από το δυναμικό του ΝΑΤΟ, να αξιοποιεί τις δυνατότητες που έχει μέσα στο ΝΑΤΟ, από το να προσπαθεί να φτιάξει ανεξάρτητες δομές. Μιλάσατε, μιλήσατε για, τις, ε, για τα battle groups της δύναμης κρούσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται όντως για μια επιχείρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φυσιολογικό είναι να μιλούμε για την ανάπτυξή τους αλλά με δεδομένη την ε, ε, ενισχυμένη δέσμευση ότι θα ήταν σε αυτές οι δυνάμεις στη Βοσνία σε περιπτώσεις όπου είναι σταθερές ε, οι συνθήκες στη Βοσνία και αυτό λέει η δική μου εμπειρία είναι λίγο δύσκολο να αναπτυχθούν. Πάντως θεωρώ ότι εάν τυχόν άλλαζε η κατάσταση στη Βοσνία σημαντικά προς τα χείρο και δεν πιστεύω ότι θα συμβεί ούτε και το ελπίζω φυσικά αλλά εάν τυχόν και άλλαζε προς τα χείρο η τάση των κρατών σε σχέση με πιθανή δέσμευση πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως της προέλευσής τους, θα ήταν ασφαλώς πολύ πιο θετική. Άρα, για εμάς, που η πολιτική μας ήταν να εξασφαλίζουμε πως οι δυνάμεις κρούσεως αντιλαμβάνονται το εύρος και το είδος των επιχειρήσεων που μπορεί ενδεχομένως να χρειαστεί να αναλάβουν ώστε να είναι προετοιμασμένες κατάλληλα και καταρτισμένες και γιατί προς έχει γίνει αυτό αλλά πάντως οπωσδήποτε το ΝΑΤΟ διατηρεί δυνάμεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να υποστηρίξουν μια ευρύτερη επιχείρηση εφόσον αυτό ήταν καθίστατο απαραίτητο. Και βεβαίως, εάν προέκυπτε μίζων κλιμάκωση, τότε θα έπρεπε να κοιτάξουμε και αυτό το ενδεχόμενο που αναφέρονται. Για τον κύριο Γκάλερ, μιλήσατε για το μέγεθος της EU4 και αν είναι επαρκές, αν είναι το κατάλληλο. Δεν είναι μόνο πολιτικό, είναι και στρατιωτικό το ερώτημά σας. Εγώ θα απαντήσω σε εξής. Με 600 άντρες υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας διοικητής στην περιοχή. Και πάλι, πάλι έχει τη δυνατότητα μιας άμεσης παρέμβασης. Δώσαμε και το παράδειγμα του Μόσταρ και όλα αυτά. Εάν μειωθεί όμως σημαντικά αυτή η δύναμη, θα είναι απίστευτα δύσκολο να αναλάβουμε δράση. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε λίγο πολύ στα όρια μιας δύναμης με εκτελεστική εντολή. Εάν έφευγε η εκτελεστική εντολή, τότε αλλάζουν τα πράγματα γιατί δεν χρειάζεται να υφίστανται, να παραμένουν σε μια χώρα η οποία, ε, σε μια χώρα στην οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μεγάλες δυνάμεις. Αν αλλάζαν τα πράγματα ε, ριζικά στη Βοσνία και δεν έκανε τίποτα η Βοσνία θα ήμασταν μάλλον ε, ανεπαρκείς αν κρατούσαμε εκεί μεγάλες δυνάμεις. Άρα νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και από την εντολή και ίσως μπορεί να προβλεφθεί η μείωση, σε, η υποβάθμιση του ΣΥΠΗΝ σε ένα επιτελείο κατάρτισης περισσότερο και διοικητική εποπτεία. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε εκείνο το πεδίο. Πάντως η EU4 ε, εξακολουθεί να παρουσιάζει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη δυναμικού και την κατάρτιση. Αυτή ενισχύεται σημαντικά από τις πολιτικές δομές που υφίστανται στη Βοσνία και αν και για να μπορέσουμε να δούμε πραγματική πρόοδο στον χώρο της άμυνας αλλά και άλλους ε, τομείς της διαχείρισης, διακυβέρνησης του κράτους θα χρειαστεί ασφαλώς να γίνουν κάποιες αλλαγές στις υφιστάμενες δομές. Αλλά βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο θα κρυθεί στο πολιτικό πεδίο. Παρατήρηση κάνω μόνο. Εν τω μεταξύ, η U4 συνεχίζει με την ανάπτυξη δυναμικού και κατάρτιση διατήρει τις δυνάμεις της, περιορισμένη δυνατότητα παρέμβασης, είναι εξτρέμις. Εφόσον βέβαια οι ένοπλες δυνάμεις της ίδιας της Βοσνίας και Ζεγοβίνης δεν είναι σε θέση να αναλάβουν δράση. Είτε απαγορεύεται είτε δηλαδή είναι ανάρμοστο. Με τα όσα είδαμε τον προηγούμενο Φεβρουάριο και το δυναμικό βίας που υφίσταται η διατήρηση μιας ε, μονάδας τέτοιου μεγέθους με εκτελεστική εξουσία, με εκτελεστική εντολή είναι σοφή επιλογή και θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις Φωσνίας και Ερσεγοβίνη είναι από τους λίγους εθνικούς θεσμούς που φαίνεται να συνενώνουν τις αντιπαλώμενες πλευρές μέσα σε μια διαδικασία αναδιάρθρωσης ε, και βλέπουμε ότι έχουμε κάνει μια οργάνωση η οποία είναι υπερήφανη για αυτό που κάνει, σεμνύνεται για τον ρόλο της, το βλέπουμε αυτό σε κάθε είδους τελετή που έχουμε παρακολουθήσει και άλλωστε αντικατοπτρίζεται και στις παρεμβάσεις, είτε πρόκειται για το Αφγανιστάν, είτε πρόκειται για υποστήριξη σε ανάγκες για πολιτική προστασία όπως οι πλημμύρες που είδαμε πέρσι. Σε αυτά όλα νομίζω ότι μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ στρατηγέ. που ήρθατε να μας μιλήσετε. Ευχαριστούμε σας προσωπικά. Ευχαριστούμε και την EU4 και την Αποστολή Αλθέα που έρχεται και μας ενημερώνει στην Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Άμυνα. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και για τις πληροφορίες. Παρακαλώ ένα μικρό ε, διάλειμμα για να ξαναρχίσουμε το επόμενο θέμα. and Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε πολύ απαιτητική ημερήσια διάταξη σήμερα. Μετά την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον στρατηγό Μπράτσο, έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Θα ήθελα να καλωσορίσω εγκάρδια τον πρέσβη Κωνσταντίνη Λισέγεφ, που είναι επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Του ζητήσαμε να μας κάνει μια σύντομη επισκόπηση της ε, στρατηγικής, πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες ε, επιθέσεις και βομβαρδισμό στο, στη Μαριούπολη. Και <clears throat> μετά την παρουσίαση της, των προτεραιοτήτων της Λετωνικής Προεδρίας, ο υπουργό Εξωτερικών της ε, Λετωνίας μας ενημέρωσε στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την παρουσία ε, του Νατοϊκού Κέντρου Αριστείας για τι στρατηγικές επικοινωνίες και τις νέες ε, αρμοδιότητες. Και θα ήθελα να καλωσορίσω τον πρέσβη Γιάννη Σκάκλινς που είναι διευθυντής αυτού του νέου κέντρου αριστείας του ΝΑΤΟ. Είναι ένας πολύπειρος διπλωμάτης και οι επιχειρήσεις και δραστηριότητες του κέντρου αριστείας του ΝΑΤΟ στη Ρήγα ε, συνδέονται άμεσα με την κατάσταση στην Ουκρανία και την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τη ρωσική επίθεση. Και ο κύριος Πρέσβης θα μας κάνει μια γενική παρουσίαση των ε, δραστηριοτήτων του Κέντρου Αριστείας και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένα σχέδια που δρομολογούνται. Ε, κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο πρώτα, κύριε Λισέγεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Φωτίγκα, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση προκειμένου να ενημερώσω την Επιτροπή σας, την σας σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες, η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα τεταμένη και απρόβλεπτη. Η Ρωσία ενίσχυσε τις αθέμητες και παράνομες δραστηριότητες της και τις διμε... αθέτησε τις διμερείς τις υποχρεώσεις και τις πρόσφατες δεσμεύσεις που έλαβε με βάση τη Συμφωνία του Μίνσκ. Γνωρίζετε ότι από την αρχή της ε, επίθεσης ε, πέρυσι το Φεβρουάριο η ε, Ρωσία συνεχίζει να κατακλείζει το ουκρανικό έδαφος με εξεζητημένο στρατιωτικό εξοπλισμό και προσωπικό και στρατιώτες και φαίνεται ότι έχουμε 40.000 περίπου στρατιωτική δύναμη στην περιοχή 8.500 ε, εκ των οποίων είναι Ρώσοι στρατιώτες ε, από τακτικά στρατεύματα της Ρωσίας και το τονίζω αυτό. Ξέρετε ότι με βάση πληροφορίες που έχουμε η Ρωσία έχει ε, φέρει στον Ντομπάς ε, στη, στη, και στις περιοχές του Ανέφ και Λουγκάνσκ παράνομα πάνω από 500 τεθωρακισμένα, πάνω από 500, πάνω από 500 συστήματα πυροβολικού και πολύ εκλεπτισμένα συστήματα εκτοξευτήρων, ε, ρουκετών και πυράβλων. Ουσιαστικά η κοιλάδα του Ντομπάς έχει γίνει ένα πολύγωνο εξάσκησης του εξεζητημένου στρατιωτικού εξοπλισμού της Ρωσίας. Τις τελευταίες μάλιστα εβδομάδες η Ρωσία ενίσχυσε αυτές τις ανατρεπτικές της επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας και έχουμε πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι αυτή τη στιγμή η Ρωσία ε, ενισχύει και τρομοκρατικέ ενέργειες σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Πρόσφατα είχαμε τρομοκρατικέ ενέργειες στην κεντρική Ουκρανία και σε νότιε πόλει, όπω το Μικολάιεφ και επίσης ε, οι μυστικές μας υπηρεσίες συγκέντρωσαν στοιχεία ότι τέτοιου είδους ανατρεπτικές ε, τρομοκρατικές ενέργειες ε, οργανώθηκαν, σχεδιάστηκαν και ενορχιστρώθηκαν από τη γειτονική μας χώρα. Μάλιστα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και ένα νέο φαινόμενο. Η Ρωσία άλλαξε την τακτική της και φαίνεται ότι εξάγει και τρομοκρατία προς την Ουκρανία. Είναι ε, να αναφέρουμε και την περίπτωση Μαριούπολης ε, και βομβαρδίστηκε περιοχή με άμαχο πληθυσμό και μάλιστα στην ε, ανατολική περιοχή της Μαριούπολ ε, βομβαρδίστηκε μια συνοικία και ε, με 12.000 κατοίκους. Στη Μαριούπολη έχουμε και σημαντική ελληνική μειονότητα και με βάση τις ουκρανικές στατιστικές πληροφορίες έχουμε περίπου 60.000 ε, Έλληνες, ε, μέλη της ελληνικής μειονότητας που διαμένουν στην Μαριούπολη και μάλιστα πριν από ε, δύο μέρες είναι περίπου που η Ελλάδα φαίνεται ότι μπλόκαρε την ενίσχυση των, κυρώσεων προς τη Ρωσία. Ενώ η βασική μειονότητα που πλήγεται στη Μαριούπολη από τους βομβαρδισμούς είναι ελληνική. Είναι πολύ περίεργη αυτή η μεταστροφή της Ελλάδος ε, και δεν ξέρω ποια θα είναι ε, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπόν κρατών μελών. Μάλιστα και η Ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης της ΟΑΣΕ συγκέντρωσε στοιχεία που ε, δείχνουν ότι η Μαριούπολη βομβαρδίστηκε από ε, αυτονομιστές, από ρωσόφιλους ε, αυτονομιστές και στόχος ε, των ενεργειών αυτών είναι ο εκφοβισμός του άμαχου πληθυσμού. Και μάλιστα ο εκφοβισμός, η τρομοκράτηση ουσιαστικά του άμαχου πληθυσμού της Μαριούπολης είναι δυνατή επειδή συνεχίζεται η απρόσκοπτη ροή στρατιωτικού εξοπλισμού και μισθοφόρων από τη Ρωσική Ομοσπονδία προς την Ανατολική Ουκρανία. Και το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να γίνει είναι να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός έλεγχος των ρωσοκρανικών σύνορων με επιτήρηση δυνατών του ΟΑΣΕ. Είναι εκ των όνων κάνευ προϋπόθεση για οποιαδήποτε σταθεροποίηση και αποκλιμάκωση της κατάστασης στις περιοχές του Ντονέτς και του Λουγκάνσκ. Επίσης, έχουμε ταυτόχρονα πολλά προβλήματα λόγω της ανθρωπιστικής κατάστασης που δημιουργήθηκε. Η Ρωσία φαίνεται ότι ετοιμάζει μια ακόμη εντός εισαγωγικών ανθρωπιστική πομπή που θα στείλει προκειμένου να στηρίξει τους ε, τρομοκράτες που χρηματοδοτεί. Και επιπλέον θα ήθελα να απευθύνω και πάλι έκκληση στη Ρωσία να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις υποτιθέμενες ανθρωπιστικές πομπές για να στέλνει πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό σε τρομοκράτες που εξακολουθούν να υπονομεύουν και να υποσκάπτουν την εδαφική αικαιρεότητα και τη σταθερότητα στην Ουκρανία. Επίσης, παρά τις προκλήσεις της Ρωσίας, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι στρατευμένη και προσιλωμένη στην ανάγκη ειρηνευτικής επίλυσης της παρούσας κατάστασης, γιατί η ειρήνη είναι η μόνη λύση στην περιοχή και στην Ουκρανία αλλά και στην Ευρώπη. Η ειρήνη είναι η μοναδική λύση. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια πρόσφατη επιστολή που έστειλε πριν από δύο μέρες ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Ποροσέγκο, προς τον πρόεδρο Πούτιν. Ο πρόεδρος Ποροσέγκο ζητά στην επιστολή του από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να εφαρμόσει πάρα αυτά και τα 12 σημεία της συμφωνίας του Μίνσκ. Και τα 12 σημεία, το υπογραμμίζω. Δεν πρέπει να διαλέγει όποια σημεία τον βολεύουν, να εφαρμόσει ολόκληρη την ε, συμφωνία του Μίνσκ και ζήτησε επίσης από τη ρωσική ε, πλευρά να σταματήσει την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού στους ε, ρωσόφιλους ε, τρομοκράτες και να καθίσει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Και μάλιστα και ο πρόεδρο Προσέγκο συνεχίζει τις επαφές του με, με Ευρωπαίους ηγέτες. Είχε χθε πολύ έντονες, διαπραγματεύσει και με τον πρόεδρο της ε, Γαλλία και με την καγκελάριο Μέρκελ προκειμένου να συγκληθεί νέα διάσκεψη υψηλού επίπεδου με θέμα την ε, επίλυση της κατάστασης με ειρηνευτικό τρόπο και την αποκατάσταση της σταθερότητας στο Λουγκάς και το Νέτσκ. Η ανθρωπιστική κατάσταση, όπως σας είπα, επιδεινώνεται η ανθρωπιστική κρίση ε, πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν ε, μετατοπιστεί εσωτερικά και η Ουκρανική κυβέρνηση έχει αναλάβει άνευ προηγουμένου προσπάθειες για να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια πρόκληση της ανθρωπιστικής κρίσης. Οι Ουκρανικές αρχές ε, συνεχίζουν να παρέχουν ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο στις κατεχόμενες από τους τρομοκράτες περιοχές και Καθημερινά δίνουμε 10 με 15 χιλιάδες κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην περιοχή Δονέτς και Λουγκάνσκ και μηνιαίως δίνουμε πάνω από 500 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και μάλιστα δωρεάν φυσικό αέριο προς το Λουγκάνσκ και τον Ντονέτσκ. Δεν λαμβάνουμε καμία αμοιβή γι' αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε τις συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα στους κατοίκους των κατεχόμενων περιοχών. Γιατί είναι και Ουκρανοί πολίτες και θα πρέπει να τους φροντίσουμε. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την ευγνωμοσύνη μου προς εσάς αγαπητοί φίλοι για τη βοήθεια και τη συνδρομή σας για τη βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Ουκρανία. Χάρη στο πρόσφατο σας ψήφισμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να δραστηριοποιείται καλύτερα και ο κύριος Τηλιανίδης πρόσφατα έρθει στην Ουκρανία, ο αρμόδιος επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια και οργάνωσε και συντόνισε μια πολύ σημαντική ανθρωπιστική πομπή στην περιοχή και χάρη στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ε, να αυξήσει την ε, οικονομική στήριξη για να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κατάσταση. ήταν πρωτοφανής αυτή η πρόβλεψη επιπλέον 15 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Συνδρομή ε, στην Ουκρανία έρχεται σε 92 με 95 εκατομμύρια ευρώ. Και πάλι θερμά ευχαριστώ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση που έδειξε στον Ουκρανικό λαό σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της Ουκρανικής ιστορίας. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι και είμαι στη διάθεσή σας ε, για να απαντήσω σε απορίες σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη, κύριε και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Πρέσβη Γιάννης Κάρκλινς για να παρουσιάσει τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ του Κέντρου Αριστείας Στρατηγικής Επικοινωνίας. Να μας παρουσιάσει λοιπόν τα έργα του κέντρου αυτή. Θα του ζητήσω λοιπόν να πάρει το λόγο και θα ζητήσω από τους βουλευτές να σχολιάσουν και τα δύο σημεία και τις δύο παρεμβάσεις ε, στη συνέχεια στο γύρο απαντήσεων γιατί έχουμε και μια πολύ σημαντική ακρόαση στη συνεδρίαση τη σημερινή. Σήμερα το πρωί θα πρέπει να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί γίνεται. Διαδικαστικό κύριο Γκάλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω, όπω είπατε δικαίω, και τα δύο θέματα είναι συνδεδεμένα μεν, αλλά αξίζουν, θεωρώ, ξεχωριστή εξέταση. Νομίζω ότι το πεδίο του κυρίου Κάκλιντ, παρά το γεγονός ότι συνδέεται με την σημερινή κατάσταση, είναι πολύ πιο ευρύ. Εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να κάνουμε έναν μικρό γύρο ερωταπαντήσεων με τον πρώτο πρέσβη και μετά να ακούσουμε τον κύριο Κάρκλινς. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ιδάλλως θα βρετευτούμε. Κύριε Φαμπάλεν, σύμφωνα με τον κύριο Γκάλερ, να είναι συγκεκριμένε οι ερωτήσει μας. Καλύτερα να ξεκινήσουμε με τον ε, πρώτο πρέσβη, λοιπόν. Εκτό μικροφώνου η Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Γκάλεφ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν συντομία κύριε πρέσβη. Χαιρόμαστε που βρίσκεστε εδώ και είμαστε ευγνώμονε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είμαστε και εμεί ε, ορατοί στην Ουκρανία σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Είμαι βέβαιος ότι τα ανθρωπιστικά μας, οι ανθρωπιστικές μας αποστολές περιλαμβάνουν σε σχετικά τρόφιμα και ό,τι χρειάζεται ο κόσμος. Μία ερώτηση για την παρουσία του ΑΣΑ και αυτά που λένε σε ό,τι αφορά τη Μαριόπολη. Θα πρέπει να είμαστε σαφείς από πού προήλθε. Σε κάποιες περιπτώσεις έχω την εντύπωση ότι βλέπουμε διάφορες ε, ενδείξεις στο facebook, στο ίντερνετ για μια σαφή παρουσία ρωσική στην μας. Σύμφωνα με τις δικές σας εκτιμήσεις, για ποιο λόγο ο ΑΣΑ πλοκάρεται λόγω της ομοφωνίας που χρειάζεται, λόγω της Ρωσίας, λόγω αυτά, αυτών που λέει, ή μήπως δεν έχει επαρκή άτομα επιτόπου για να δώσει τα δεκμήρια που χρειάζονται. Ευχαριστώ κύριε Σατίνα. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Συχνά τον τελευταίο καιρό ρωτώ τι είναι πιο σημαντικό σε αυτή τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Είναι άραγε η τόνοι πυρομαχικών, τάγκς ή τόνη λέξεων. Και αυτό το ρωτάω για τον εξή λόγο. Γιατί βλέπουμε ότι σίγουρα γίνεται και ένας πόλεμος πληροφοριών εδώ. Και αυτό κινείται μάλλον προς όφελος των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας, γιατί τα ψέματα ως εργαλείο πολιτικής του Κρεμλίνου και ως εργαλείο της ρωσικής διπλωματίας, ας μην ξεχνάμε την διπλωματική σχολή που ακόμα θεωρεί τα ψέματα διπλωματικό εργαλείο. Να ρωτήσω λοιπόν τη γνώμη σας, κύριε Πρέσβη, τι κάνει η Ουκρανία για να καταπολεμήσει αυτή τη μεγάλη εισρωή ψευδών δηλώσεων στην πολιτική σκηνή και στα μέσα ενημέρωση. Και υπάρχουν κοινά μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Μαρέκ Γιούρεκ, λέει πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Όλοι παρακολουθούμε την κατάσταση στην κοιλάδα του Ντονέτσκ, στον Ντομπάς. Και είπαμε και πολλές φορές ότι αυτή η τραγωδία στην Ουκρανία δεν θα δημιουργήσει συγκεκριμένες ε, τάσεις. Ε, είχαμε δύο βομβαρδισμούς ε, αμάχων στον Ντονέτσκ, τώρα έχουμε τέτοιο βομβαρδισμό και στη Μαριούπολη. Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση όμως ε, για την ασφάλεια και την εξάπλωση της σύγκρουσης ε, σε δύο άλλες ε, περιοχές. Τι κάνει η Ρωσία στην Κρυμαία, έχετε στοιχεία για ενέργειες της Ρωσίας εκεί. Επίσης, τι γίνεται στο Δνιέστρε, παρακαλώ ολοκληρώστε, τι γίνεται στην Οδυσσό και την ασφάλεια της Οδυσσού. Κύριος Βανβάλεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη έχουν καταδικάσει τόσες πολιτικές ομάδες της, ε, τη δράση της Ρωσίας και ζητούν επιπλέον κυρώσεις σήμερα. Όχι μόνο εγώ αλλά και άλλοι εδώ. Από τη στρατιωτική όμως ε, θεώρηση, μια και είμαστε στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, θέλω να ρωτήσω εάν η Ουκρανία έχει δυνατότητα, δυναμικό για να κρατήσει τους Ρώσους έξω από τη Μαριούπολη. Δεν είμαστε σε συνεδρίαση και των θυρών και έτσι ξέρετε ότι δεν μπορείτε να δώσετε διεξοδική απάντηση αλλά έχετε τη δυνατότητα, έχετε τη στρατιωτική ικανότητα να βοηθήσετε σε αυτή την πτυχή των κυρώσεων. Ο κύριος Ζέμκε, εγώ θα ήθελα να συνεχίσω τις ερωτήσεις του συναδέλφου γιατί εμεί είμαστε υπό Επιτροπή ασφάλειας και άμυνας. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω όχι μόνο για το δυναμικό, γιατί από τις 11 Σεπτεμβρίου άρχισαν οι μάχες και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις είναι μάλλον ζωφερές οι προοπτικές. Τι, τι δυνατότητα εξοπλισμού ε, έχει αυτή τη στιγμή ο Ουκρανικός στρατός. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαντσπέρκης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλημέρα σας, με χαρά σας βλέπουμε εδώ στο κοινοβούλιο, κύριε Ελισέγεφ. Ε, η εικόνα πρέπει να είναι απόλυτα σαφής όταν μιλούμε για τα θέματα της προσέγγισης με τη Ρωσία ή την ε, παραβίαση των συνόρων. Θα πρέπει να καταστεί σαφέ δηλαδή ότι ακόμα και δύο εκατοστά παραπάνω να προχωρήσουν θα έχουν πιο σοβαρέ κυρώσει να αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, είχαμε την υπογραφή της συμφωνίας με την ε, Ουκρανία για μια πιο εκτεταμένη αμυντική συνεργασία. Μπορείτε να εξηγήσετε τι περιμένετε, τι, σε τι μπορούν να συμβάλλουν τα άλλα κράτη, πού μπορείτε να ζητήσετε περισσότερη βοήθεια και τι θα μπορούσαμε εμείς να προσφέρουμε επί τη ευκαιρία του παραδείγματος αυτού. Και κάτι ακόμη, μπορείτε να μας κάνετε να μας ξαναδείξετε την κατάσταση, να μας εξηγήσετε πάλι την κατάσταση για την κινητοποίηση, γιατί ε, υπόθηκε ότι έχει ανακοινωθεί μια μερική επιστράτευση. Μπορείτε λοιπόν να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες και εάν υπάρχουν νεκροί Ρώσοι στρατιώτες στην Ουκρανία, στρατιώτες στην Ουκρανία, πώς το αντιμετωπίζετε το θέμα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος. Θέλω λοιπόν αποδείξεις. Γιατί μας μιλήσατε για εισβολή. Μα δείξετε όμω το δορυφόρο μια εμπορική εταιρεία. Πού είναι οι αποδείξεις ε, για, για την παρουσία Ρώσων στρατιωτών στην περιοχή ή για τη χρήση Τρομοκρατία. Πού είναι οι αποδείξει, πού είναι τα τεκμήρια. Επίσης, ε, Μιλήσατε για εκτοξευτήρες ε, πολύ σύγχρονου και εκλεπτισμένου. Τι, τι συνέβη με τη Μαριούπολη, το ίδιο με το Μαλαισιανό αεροσκάφο. Ακόμη δεν βρήκαμε τον ένοχο. Γιατί διαταράχθηκε η ανακοχή. 22 Ιανουαρίου οι Ουκρανοί ε, επιστέθηκαν στο Ντονέτσκ. Είχαμε 13 με 15 νεκρούς στο Σταχάνοβο μετά από λίγες μέρες. Ε, είχαμε 8 νεκρούς, 2 παιδιά. Ε, την περασμένη εβδομάδα συνέβη κάτι τέτοιο και καμία καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ας αφήσουμε τη, τις, παθιασμένες ομιλίες και να βρούμε ε, μία ε, λύση ειρηνευτική για να προστατεύσουμε τον άμαχο πληθυσμό. Ο κύριος... Ευχαριστώ κύριο Σκέλαμ και κλείνω ο κατάλογος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρέσβη. Για να απαντήσω στον προλαλήσαντα που ρωτούσε που βρίσκονται οι αποδείξεις. 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα της ε, Εσθονίας υπάρχει η μεραρχία Σκόπ στρατιώτες και αξιωματικοί από αυτή τη μεραρχία, σε απόσταση μεγάλη από την Ουκρανία, έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω σε επιχειρήσεις και έχουν ε, ταφεί στο σκόπ. Νομίζω υπάρχει δυνατότητα να προληφθούν τέτοιου είδου επιθέσει. Υπήρχε ήδη μια εβδομάδα νωρίτερα ένδειξη σαφή, ότι ενισχύουν οι Ρώσοι την παρουσία του στα σύνορα. Όλα τα δεδομένα έδειχναν ότι ετοιμάζουν επίθεση. Θεωρείτε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα έπρεπε προληπτικά να δράσουν για να αποφύγουμε τέτοιου είδου επιθέσει. Ο πρέσβης Ηλισέγεφ παρακαλώ για να απαντήσει και να δώσει παρατηρήσεις του. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας και για τις σημαντικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Για τις δραστηριότητες καταρχάς και την αποστολή όσα ο ΑΣΕ. Ναι βεβαίως και, και θα είναι χρήσιμη. Πολύ σωστά λέτε ότι δρά με βάση συνενετική. Ταυτόχρονα, ξέρετε, η αποστολή ο στην Ουκρανία παρουσιάζει καθημερινά τις εκθέσεις της στα γραφεία στη Βιέννη και αν διαβάζετε τις εκθέσεις αυτές θα βλέπατε ότι υπάρχει σαφέστατη κινητοποίηση βαρέως εξοπλισμού και δυνάμεων βεβαίως χωρίς ε, τα χαρακτηριστικά σύμβολα ε, αλλά πάντως κινητοποίηση κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας. Και θέλω να πω ότι όταν μιλούμε για την αστροειδική παρουσία της Ρωσίας και της ρωτικά στρατεύματα πριν μπουν στα εδάφη της Ουκρανίας παίρνουν οδηγίε να ξέρετε όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες να βγάλουν όλα τα χαρακτηριστικά, όλα τα ε, στοιχεία που έχει στολή για τον εντοπισμό και κάθε είδους στοιχείο ταυτότητας ή έγγραφο που θα μπορούσε να τους ταυτοποιήσει. Άρα εμείς σταριζόμαστε περισσότερο στην ε, τέχνογνωσία, την ε, εμπειρία και τη βοήθεια τεχνική που μπορεί να μας προσφέρει ο ΑΣΕ. Από αυτούς έχουμε σαφείς ενδείξεις και έγγραφα που δείχνουν ότι υπάρχει κινητοποίηση ρωσικών στρατευμάτων. Επίσης, δεν εντείνονται οι, δεν εντείνονται οι εγγύσεις για την ασφάλεια του προσωπικού του ΑΣΕ από πλευράς των τρομοκρατών οι οποίοι δεν δέχονται να επεκτείνουν την προστασία του προσωπικού αυτού στις περιοχές που ελέγχουν. Αλλά ας περάσω πάλι στη Μαριούπολη. Την τρομοκρατική επίθεση στη Μαριούπολη και αγαπητοί φίλοι, σας έχω αποστείλει κάθε υλικό ε, καταγραφής κινήσεων που έχουμε από την ε, μυστική υπηρεσία της Ουκρανίας για να αποδείξουμε ότι έχει οργανωθεί από τη στρατηγική διοίκηση της Ρωσίας και με τη βοήθεια της, ε, των Ρώσων τρομοκρατών αυτή η επίθεση. Γιατί σταμάτησαν, γιατί άρχισαν ε, να κυκλοφορούν οι καλές ειδήσει ότι πάνε οι παρατηρητές του ΟΑΣΕ να δουν τι συμβαίνει στη Μαριούπολη. Μόλις κυκλοφόρησε αυτή η είδηση, αμέσως εδόθη η εντολή να αποσυρθούν τα συστήματα ρήψης πυράβλων και όλα τα άλλα ρωσικά συστήματα για να μην μπορούν να αναγνωριστούν ως ρωσικά. Πυροβολικό, αν δείτε το υλικό που σας στέλνω, θα διαπιστώσετε ότι μπορέσαμε να συλλάβουμε κιόλας κάποιον. Συντονιστή μάλιστα, ο οποίος δηλώνει ξεκάθαρα ότι όλα αυτά τα έχει ετοιμάσει και οργανώσει η ρωσική στρατιωτική διοίκηση. τα ψέματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η προσπάθεια για την ε, α, κατάρριψη των ψευδών επιχειρημάτων της ρωσικής προπαγάνδας. Αυτός είναι ο μεγάλος μας αγώνας. Ξέρετε, πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση για τις Ουκρανικές αρχές και την κυβέρνησή μας είναι να καθαρίσουμε τις ε, νοοτροπίες και τις ε, προτιμήσεις θα έλεγα των ανθρώπων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές γιατί οι ρωσικές αυτές δυνάμεις, ρωσόφιλες δυνάμεις στηρίζονται στην ε, υποστήριξη τοπικού πληθυσμού. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει ε, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ουκρανική, ακόμα και ίντερνετ, δίκτυα κοινωνικής επικοινωνίας, και η μόνη επικοινωνία που έχουν ε, με τον έξω κόσμο προέρχεται από την επαφή την, από την παρακολούθηση της ρωσικής τηλεόρασης αλλά βέβαια έχουμε ένα έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων σήμερα το οποίο θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Επίσης, ένας άλλος ε, ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στη στρατική υποστήριξη και τις ελλείψεις στον Ουκρανικό στρατό. Πολύ σωστά αναφέρατε ότι είναι ε, ευαίσθητο ζήτημα και δεν μπορώ να εκθέσω πολλές λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία ακόμη και από εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά και στις 28 χώρες μέλη, εργάζεται εντατικά ε, για να ζητήσει περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη και εδώ και βέβαια στο Συμβούλιο για να εξασφαλίσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την ε, ενθάρρυνση των κρατών μελών για περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας στο πλαίσιο βεβαίως των εφισταμένων νομικών διατάξεων, νομοθετικών διατάξεων. Αυτή την υποστήριξη ζητούμε. Γιατί μέχρι στιγμής μόνο μη φωνικά όπλα όπως ονομάζονται, non-lethal weapons, μπορούμε να λαμβάνουμε. Εμείς χρειαζόμαστε όμως κάθε τύπου στρατιωτική υποστήριξη. Και πάλι όπως είπα, τα κράτη-μέλη με τα οποία έχουμε επικοινωνία ξέρουν πολύ καλά ποιες είναι ανάγκες μας και τι μπορούν να μας προσφέρουν. Στο θέμα λοιπόν αυτό για τη Μαριούπολη η Ουκρανία κατάφερε να υπερασπιστεί τη Μαριούπολη. Ναι, μπορέσαμε να υπερασπιστούμε τη Μαριούπολη. Με τη βοήθεια και του τόπιου πληθυσμού, πρέπει να πω, μπορέσαμε να στήσουμε τρεις αμετικές γραμμές και σας διαβεβαιώ, αγαπητοί φίλοι. Εάν μπορέσουν να επιστρέψουν οι Ρώσοι τρομοκράτες στη Μαριούπολη, θα γίνει σφαγή εκατόμβη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν για να την υπερασπιστούμε. Σε σχέση με τους ρόστρατιώτε που ενδεχομένω έχουν σκοτωθεί. Θα σα πω ένα γεγονό. το ανακαλύψαμε χθε. Μια-δύο εβδομάδε πριν ανακαλύψαμε είχε αναπτύξει ένα κινητό κρεματόριο η Ρωσία. Έχουμε πραγματικά στοιχεία, γεγονότα. Απάνθρωπο βέβαια αυτό. Γιατί ξέρετε εμείς στη Ρωσία όλο και πιο πολλές ε, εκκλήσεις λαμβάνουμε από μητέρες, πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας που μας ζητούν τη βοήθειά μας για να ξαναβρούν τα παιδιά τους, ε, κορίτσια, αγόρια τους, συζύγους τους, τα αδέλφια τους αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να την αναλύσουμε από την ανθρωπιστική βέβαια ε, προοπτική. Και επίσης θέλω να αναφερθώ στα στοιχεία για άλλη μια φορά που έχουμε, τα αποδεικτικά. Εγώ όπως είπα, έχω στη θέση μου στοιχεία, μπορώ να σας διαθέσω προσωπικώς, προερχόμενα από διάφορε πηγέ. Αν όμω δεν σα φαίνονται πιστεπτά τα, τα, κριτήρια, τα πιστήρια τη Ουκρανία, κοιτάξτε παρακαλώ προσεκτικά τι εκθέσει του ΟΑΣΕ, που όμω και πάλι έχουν ε, προβλήματα. Ξέρετε, δεν μπορεί να αναπτύξει μη επανθρωμένα αεροπλάνα, γιατί οι Ρώσοι έχουν στη δυνατότητά του ε, ε, εξοπλισμό, ο οποίος μπορεί να, παρε... να κάνει παράσιτα στη λειτουργία αυτών των αεροπλάνων και άρα δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Και για τον κύριο Κέλαμ, και τις ερωτήσεις του. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να πολεμήσουμε μόνοι μας. Φυσικά χρειαζόμαστε στρατιωτική ε, και τεχνική υποστήριξη από άλλες χώρες. Εμείς δεν θέλουμε να μας στείλετε δυνάμεις ενόπλες ε, από γειτονικά ή άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ξέρετε ότι έχει καταγγείλει πρόσφατα ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ότι υπάρχει μια λεγεώνα ε, του ΝΑΤΟ ε, στην ε, περιοχή. Εμείς είμαστε θέση να επιστρατεύσουμε έως και 30.000 στρατιώτες. Ε, αυτό μας αρκεί προς το παρόν. Παρά τις διαμαρτυρίες της ρωσικής ηγεσίας ότι η Ουκρανία προσπαθεί να ενισχύσει στρατιωτική τη παρουσία και να κοινοτοποιήσει, να επιστρατεύσει πολίτε. Κοιτάξτε, αυτό είναι δικαίωμά μα. Δικαίωμα από τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την αυτοάμυνα, αγαπητοί φίλοι. Και σα διαβεβαιώνω ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ε, χώρα μα, ταυτόχρονα ελπίζοντα στην υποστήριξη και βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα. Γιατί αγωνιζόμαστε για την ελευθερία και τι ευρωπαϊκέ αξίε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ λυπάμαι που πρέπει να περιορίσω τη συζήτηση αυτή, αλλά το σημείο αυτό είναι κατεπήγον και πολύ απλά προσθέθηκε ανάμεσα στα προβλεπόμενα πολύ σημαντικά σημεία της ημερήσιας διάταξης, αλλά είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον πρέσβη Γιλτσεφ που μπόρεσε να παραστεί εδώ και να μας μιλήσει. Αν θέλετε ασφαλώς να μείνετε στην αίθουσα. Και το λόγο έχει τώρα ο Πρέσβης Κάρκλινς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να παρουσιάσω το κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ για τις στρατηγικές επικοινωνίες. Η πρωτοβουλία η οποία ξεκίνησε από την Λατινική Προεδρία για αντίδραση, ανταπόκριση στην απόφαση που ελήφθησε στην Σύνοδο του 2009 μεταξύ στο, του ΝΑΤΟ, όπου αναγνωρίστηκε ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τις στρατηγικέ επικοινωνίε του. Στόχος του κέντρου είναι να παρέχει απτή συνεισφορά στην βελτίωση των ικανοτήτων στρατηγικής επικοινωνίας του ΝΑΤΟ μέσω διάφορων δραστηριοτήτων, μέσω αναλυτικής έρευνας, μέσω πολυτομεακής δέσμευσης, μέσω βελτίωσης της διαλειτουργικότητας και των ικανοτήτων και βελτιωμένης ε, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το κέντρο δημιουργήθηκε ως Λευδονικό Εθνικό Ίδρυμα τον Γενάρη του 2014 με 3 εκατομμύρια ευρώ από τη λεπτονική κυβέρνηση, όχι μόνο για το 2014, αλλά και για το 2015 και 2016. Τον Απρίλιο έλαβε χώρα η διάσκεψη ίδρυση το 2014 και 7 χώρες ε, εξέφρασαν ενδιαφέρον και δεσμεύτηκαν και κατέστησαν ιδρυτικές χώρες. Εκτός από τις τρεις ε, Βαλτικές, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Πολωνία. Αυτές οι 7 χώρες Υπέγραψαν λοιπόν τα σχετικά έγγραφα ίδρυσης ε, την 1η Ιουλίου και το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση να πιστοποιήσει το κέντρο και να το ενεργοποιήσει ως ε, στρατιωτικό σώμα του ΝΑΤΟ το Σεπτέμβριο του 2014 το κέντρο αριστείας. Ήταν το 20ο κέντρο αριστείας του ΝΑΤΟ Αποτελεί λοιπόν σώμα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν αποτελεί τμήμα της ε, δομής ε, εντολών του ΝΑΤΟ. Έχουμε μεγάλη ανεξαρτησία λοιπόν και μπορούμε να διεξαγάγουμε την έρευνά μας και την ακαδημαϊκή μας μελέτη σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες που όρισαν τα ιδρυτικά μέλη στην Διοικητική Επιτροπή. Το 2014 επίσης ξεκινήσαμε τις ουσιαστικές μας λειτουργίες και δραστηριότητες. Διεξαγάγαμε μία σειρά εκπαιδεύσεων. για τους αξιωματικούς ε, της Ουκρανίας και της ε, αξιωματικούς του κράτους. Κάναμε διάφορες έρευνες καταρχάς ε, για την πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ και σε ό,τι αφορά την περίοδο 2017 και 2013 κάναμε μία μελέτη η οποία ήταν εντολή του Λιτωνού Υπουργού Άμυνας για τις ε, εκστρατείες πληροφόρησης της Ρωσίας κατά της ε, Ουκρανίας κοιτώντας ε, την περίοδο από το Νοέμβριο του 2013 στη διάσκεψη του Βίλνιους μέχρι την προσάρτηση της Κρυμαίας το Μάρτιο του 2014. Επίσης, ε, κοιτάξαμε το πώς εξελίχθηκε η σύγκρουση από στρατηγικής απόψεις Και μετά, την περίοδο αυτή ασφαλώς, διεξάγαμε κάποια αρχικά σεμινάρια για ε, επίκαιρα ζητήματα για το πώς τα κοινωνικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο σε υβριδικό πόλεμο. Το 2015 εργαζόμαστε σε νέα, για νέα έργα τα οποία ενδιαφέρουν και απασχολούν πολλούς, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ενημερωτική εκστρατεία για τις κοινωνίες των χωρών ΝΑΤΟ. Κάνουμε επίσης επιχειρήσεις για, από πλευράς στρατηγικής επικοινωνίας που καλύπτουν όλη την επιχειρησιακή περίοδο 2013-2014 και σε ό,τι αφορά τη συγγραφή της στρατηγικής επικοινωνίας των επιχειρήσεων αυτών. Τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη έχουν να κάνουν με την έρευνα των μέσων κοινωνική δικτύωση ως εργαλείο πολέμου και επίση μία μελέτη για το πώ θα εντοπίζονται ε, έγκυρε ενδείξει, πρώιμε ενδείξει τέτοιων υβριδικών πολέμων προκειμένου να αναπτυχθούν σχετικοί δείκτε για ένα εγχειρίδιο επίση εργαζόμαστε για το πώ το ΝΑΤΟ και τα κράτη-μέλη μπορούν να προστατευτούν από τέτοιε περιπτώσει μόχλευση. Το κέντρο μας εξετάζει λοιπόν ζητήματα ποικιλόμορφα, μεγάλης ε, και ευρείας ε, κλίμακας. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι σήμερα το περιβάλλον πληροφόρησης έχει αλλάξει δραματικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς. Αν μου επιτρέπετε, εν συντομία, θα ήθελα να αναφερθώ στα πορίσματα, σε κάποια πορίσματα σε ό,τι αφορά τη ρωσική ε, εκστρατεία πληροφόρησης κατά της Ουκρανίας. Θα ήθελα ιδιαίτερο αυτό να το δούμε στο όλο συγκείμενο, στο όλο πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τον ορισμό του ευρετικού πολέμου όπως ορίστηκε από τον στρατηγό Γκεράσιμο. Θα αναφέρω κάποιες ε, από τις ε, δηλώσεις του απορίσματο, το απορίσματα του από ένα άρθρο του 2013. Παραθέτω, το στον 20ο αιώνα υπάρχει λοιπόν η τάση να υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ των ανδρών των πολέμων που δεν ακολουθούν τη συνήθη μορφή εκκίνησης. Έχουν αλλάξει σημαντικά οι πόλεμοι. Τα μη στρατιωτικά μέσα είναι όλο και πιο σημαντικά για την επίτευξη στρατιωτικών στρατηγικών στόχων και πολύ πιο αποτελεσματικά σε κάποιες περιπτώσεις σε σύγκρουση με τις ε, στρατιωτικές δυνάμεις. Και τέλος, ότι υπάρχει μία μετάβαση από τη χρήση συμβατικών μέσων στην ε, χρήση άλλων μη στρατιωτικών μέσων, μεταξύ άλλων και της εμπλοκής και της συμμετοχής ε, του κόσμου, των αμάχων. Διαβάζοντας λοιπόν το άρθρο αυτό, θυμάμαι, θυμήθηκα αυτά που μόλις μας είπε ο πρέσβης της Ουκρανίας. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία ακριβώς αυτά που περιέγραψε ως ευρωδικό Πόλεμο ο στρατηγός Γκράσιμο. Εξετάσαμε επίσης τη σύγκρουση αυτή από ιστορικής ε, σκοπιάς και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ρωσική εκστρατεία πληροφόρησης κατά της ε, Ουκρανίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πρόκειται μάλλον ένα αποτέλεσμα μιας μακρόπνοη στρατηγικής της Ρωσίας η οποία διεξαγάγεται με διαφορετική ένταση σε διαφορετικά τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης σε μία περίοδο 15 ετών, των τελευταίων 15 ετών. Οι διάφορες μέθοδοι τις οποίες παρατηρούμε περιγράφονται τα έγγραφα πολιτικής της Ρωσίας και μάλιστα από το 2007 σε μία αναθεώρηση της πολιτικής ε, της Ρωσίας το 2007 σας παραθέτω λοιπόν τι λέει το σχετικό έγγραφο. Ο βασικός μας ε, στόχος είναι να διεξαγάγουμε αποτελεσματικές εξατίες πληροφορίες, όπου υπάρχει σημαντική πρόκληση και υπονόμευση των συμφερόντων της Ρωσίας και της ε, ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Η πολιτική, πατριωτική πολιτική της Ρωσίας παίζει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερο ρόλο θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις δράσεις που διεξαγάγει η Ρωσία σήμερα στην Ουκρανία. Και η διπλωματική δραστηριότητα της Ρωσίας στους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων και των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΑΣΕ. Αυτά λοιπόν καταδεικνύουν με σαφήνεια το μακρόπνο αυτό σχεδιασμό τη μακρόπνοη αυτή στρατηγική, ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να κατανοήσουμε είναι το εξή. Από το 1999, όταν ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Πούτιν, σταδιακά ξεκίνησε να καταργεί τα στοιχεία που καταρτίζουν και συναποτελούν τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μεθενημέρωση στη Ρωσία. Σήμερα πλέον στη Ρωσία μπορούμε να μιλήσουμε για ένα κράτος που ελέγχει τα μέσα ενημέρωσης, ιδιαίτερα τα οπτικοακουστικά. Γιατί η πλειοψηφία των μεγάλων ε, τηλεοπτικών σταθμών είτε ανήκουν στο ρωσικό κράτος, είτε ανήκουν σε εταιρείε τις οποίες ε, κατέχουν ε, Ρώσοι ολιγάρχες που πρόσκενται στο Κρεμλίνο. Το μοναδικό, ο μοναδικός σταθμός ενημέρωσης που δημιουργήθηκε το 2013 και ήταν εξάρτητος, προσπαθεί απεγνωσμένο να πετύχει κάποια ακροαματικότητα. Με πάρα πολύ λίγες λοιπόν εξαιρέσεις τηλεοπτικών σταθμών και μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να αντιταχθούν στον κρατικό έλεγχο της Ρωσίας, δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για ανεξάρτητα ελεύθερα μέσα ενημέρωση της Ρωσίας. Μιλάμε για ένα μηχανισμό κρατικής προπαγάνδας, δημοσιογράφους, πράκτορες της προπαγάνδας. Επίσης, εξετάσαμε διάφορες μεθόδους ε, πληροφόρησης που χρησιμοποιούνται. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι υπάρχει η μέθοδος διάδοσης του φόβου και είδαμε με ποιους τρόπους τα μέσα προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν α, εικόνες που προκαλούν έντονα συναισθήματα για να πείσουν, για να δράσουν σε υποσυνείδητο επίπεδο στο κοινό τους. Βλέπουμε λοιπόν ε, καταφανώς παραποίηση γεγονότων και παραπλάνηση της κοινή γνώμης. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της μελέτης αυτής εξετάσαμε τι είδους ιστορίες χρησιμοποιούνται στην ρωσική τηλεόραση στις σχετικές εξατίες. Δύο ειδών ιστορίες σε ό,τι αφορά το συγκείμενο και σε ό,τι αφορά την εκστρατεία. Σε ό,τι αφορά το συγκείμενο, τις ιστορίες, τις σχετικές, θα τις αναφέρω και θα τις παραθέσω. Έχουμε το θέμα της σύγκρουσης των πολιτισμών, της αξίας της Ορθόδοξης Ρωσικής Εκκλησίας, ο ρωσικός κόσμος εν γέννη, μια άλλη ιστορία όπου η Ρωσία, η Ουκρανία και η Λευκορωσία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και υπήρχε και η ιστορία της προώθησης ε, της ιδέας της ενότητας της Ευρασίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ιστορίες της εκστρατείας, έχουμε την ε, ιστορία με ανοιχτό τέλος, ότι συνεχίζεται ο μεγάλος πατριωτικός πόλεμος, δεν έχει έχει τηθεί ακόμα ο φασισμός και το καθεξής. Και είδαμε πόσο η Ρωσία επιθυμεί να νομιμοποιήσει τις ενεργειές της, υπενθυμίζοντας ε, διάφορα νομικά και ενωμα μέσα, κατηγορώντας τις δυτικές χώρες και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της όλης εκστρατείας η Ρωσία προσπάθησε να διχάσει ή μάλλον να παρουσιάσει διχασμένες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η μελέτη η οποία λοιπόν διατίθεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Αριστείας ε, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πληροφόρηση αποτελεί ένα πανίσχυρο εργαλείο επιρροής και αποτελεί ένα κεντρικό εργαλείο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Επίσης εξετάσαμε την ταυτοποίηση, των, τον εντοπισμό των αδυναμιών και των δυνατών σημείων των εξαρτιών. Στα δυνατά σημεία συγκαταλέγονται η σωστή, ο σωστός χρονισμός η μακροπρόθεσμη προετοιμασία, η καλή εκτέλεση, καλός έλεγχος, χρήση πατριωτικών πολιτικών και η γνώση και η κατανόηση στοχευμένων ομάδων, ιδιαίτερα στην Κρυμαία και μαζική χρήση παραπλάνησης. Μία από τις μεγάλες αδυναμίες είναι το γεγονός ότι υπάρχει συνεχής διάβρωση της εξατίας παραπληροφόρησης. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει συνοχή μεταξύ των του τι λέγεται. Και είδαμε ότι η Ρωσία επίσης δεν είναι σε θέση να ελέγξει απόλυτα τα κοινωνικά μέσα. Μέσω των κοινωνικών μέσων λοιπόν, η ροή πληροφόρησης ήταν ανεξέλεγκτη. Γιατί λοιπόν είναι όλα αυτά τόσο σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη είναι στον χώρο πληροφόρηση της Ρωσίας, ο οποίος και επεκτείνεται. Η επικέντρωση την τελευταία δεκαετία ήταν κυρίως σε αυτό που η Ρωσία αποκαλεί τις κοντινές χώρες, ε, εξωτερικές χώρες. Σήμερα ο χώρος αυτός επεκτείνεται τάχιστα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων χωρών όπω η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία πιο μακριά. Ο κόσμος λοιπόν επηρεάζεται από τη ρωσική προπαγάνδα. Η Ρωσία χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο για να προβάλλει την επιρροή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις αξίες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει. Τις εκμεταλλεύεται δηλαδή στην εξαρτία προπαγάνδας. Η Ρωσία επίση χρησιμοποιεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για να καταχωρήσει τους τηλεοπτικούς σταθμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε πέντε τηλεοπτικούς σταθμού ρωσικούς καταχωρισμένους στο Λονδίνο σε μία διεύθυνση όπου υπάρχουν καταχωρισμένες και άλλες 197 ε, επιχειρήσεις. Άλλη μία στην Λετωνία, άλλος ένας τηλεοπτικός σταθμός στη Λετωνία και άλλος ένας ε, ε, στην Σουηδία. Τέλος, θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι στο τρέχον περιβάλλον μέσων ενημέρωσης, λόγω ακριβώς των διαταραχών των υπηρεσιών τεχνολογίας, είναι πολύ εύκολο να υπάρξει επιρροή και η προπαγάνδα της Ρωσίας επηρεάζει πάρα πολύ. Τα μέσα πασχίζουν να βρουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο το οποίο θα τους επιτρέπει να επιζήσουν. Δεν έχει βρεθεί όμως αυτό το μοντέλο αντίθετα με την ε, βιομηχανία της μουσικής για παράδειγμα. Άρα είναι μεγάλε οι προκλήσει και για του δημοσιογράφου και για του τηλεοπτικού σταθμού. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τι ε, δυνατότητέ μα για στρατηγική επικοινωνία. Δεν μπορούμε να αποδεθούμε σε μια δική μα προπαγάνδα για να αντιταχθούμε στη ρωσική προπαγάνδα, αλλά θα πρέπει να πούμε τη δική μα ιστορία με έναν τρόπο κατανοητό σε όλου. Και πιστεύουμε ότι οι στρατηγικέ επικοινωνίε αποτελούν ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Σα ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε, για την ευκαιρία αυτή που μου δώσατε να παρουσιάσω το κέντρο μα και να σα μιλήσω για τα πορίσματα τη πρώτη μα έρευνα σε ό,τι αφορά την ε, εκστρατεία της Ρωσίας. Thank you. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρεσβευτά, κύριε Κάκλινς. Ε, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση που μας κάνατε για το κέντρο αριστείας και φαντάζομαι και οι συνάδελφοι θα θέσουν ερωτήσεις για άλλα θέματα. Εμένα με ενδιαφέρουν τα μελλοντικά σας ερευνητικά σχέδια. Ποια είναι, υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης των προγραμμάτων σας. Προσωπικά πάντως λυπούμε ειλικρινά για το ότι καθυστέρησε τόσο πολύ να τεθεί σε ισχύ αυτό το κέντρο αριστείας και να αναλάβει ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η ρωσική προπαγάνδα. Αν είχε αρχίσει να λειτουργεί πιο νωρίς το κέντρο αριστείας, θα είχαμε αποφύγει πολλά τέτοια θέματα. Ο κύριος Τέτινα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μία πολύ σύντομη ερώτηση. Γνωρίζω ότι οι ραδιοφωνικές εκπομπές της, ε, του ουκρανικού ραδιοφωνικού σταθμού Free Europe ε, από την Πράγα ακούγεται πολύ στην Ουκρανία. Θα ξεκινήσετε και άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς ή θα χρησιμοποιήσετε δορυφόρους για την αναμετάδοση και άλλων ε, διεθνών τηλεοπτικών σταθμών στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρεκ Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εξονυχιστική αυτή η ενημέρωση, κύριε Πρέσβη. Μήπως και μέσω άλλων ερευνητικών ε, Ινστιτούτων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσετε το θέμα της εξήμνησης του κομμουνισμού στη Ρωσία, γιατί πραγματικά η Ρωσία συνδέει την εξήμνηση του σταλινισμού ε, ε, με την προσπάθεια την αντίστοιχη που γίνεται στη Λευκορωσία γιατί η εξήμνηση του κομμουνισμού και του σοβιετικού παρελθόντος είναι κάτι που εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. Θα συνεργαστείτε με άλλα ερευνητικά κέντρα για να λάβετε υπόψη και το θέμα αυτό. Κύριε Κάκλης, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά μας σχέδια, σας έδωσα το πρόγραμμά μας για το 2015. Αρχίζουμε τώρα να σκεφτόμαστε τις αδερές γραμμές και του προγράμματος του 2016. Πάντως, ό,τι αφορά τις μεθόδους επικοινωνίας του ΙΣΙΛ, του Ισλαμικού κράτους ε, και το πώς στρατολογούν τους ξένους μαχητές από τη Δυτική Ευρώπη ή πώς οι πληροφορίες τους επηρεάζουν την κοινή γνώμη στη Δυτική Ευρώπη Επίσης, εξετάζουμε εμπειρίες από στρατηγικές επικοινωνίες από τις επιχειρήσεις της ISAF στο Αφγανιστάν για την περίοδο 2003 με 2014. Εξετάζουμε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς χρησιμοποιούνται σε υβριδικό πόλεμο. Γιατί τα αποτελέσματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ε, δεν έχουν γίνει πλήρως αντιληπτά. Επίσης, προσπαθούμε να μετριάσουμε τη χρήση των μέσων κοινωνική δικτύωσης από τους αντιπάλους μας. Άλλα σημαντικά ερευνητικά προγράμματα που θα στηρίξουμε είναι προγράμματα για να αντιληφθούμε καλύτερα το ρόλο των στρατηγικών επικοινωνιών για να εντοπίσουμε εγκαίρως και σχετικά νωρίς πιθανές επιχειρήσεις κατά μελών του ΝΑΤΟ. Επίσης, μας ενδιαφέρει και το παιδαγωγικό σκέλος ε, και θα υποβάλουμε και ένα διαδικτυακό μάθημα για στρατηγικές επικοινωνίες. Ένα διαδικτυακό σεμινάριο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κάποιες προσπάθειες και δραστηριότητες για να δούμε κατά πόσο η δημιουργία ενό τηλεοπτικού σταθμού που θα εκπέμπει στα ρωσικά θα ήταν χρήσιμη. Γίνεται τώρα μια μελέτη σκοπιμότητας ε, ενός τέτοιου σταθμού. Θα δούμε ποια θα είναι τα πορίσματά της και αν θα υποδοθεί η προσπάθεια. Ξέρω ότι η Εστονία πρόσφατα έχει εγκαινιάσει ένα τέτοιο ρωσόφωνο κανάλι ραδιοφωνικό και θα γίνουν άλλες προσπάθειες τέτοιες και αλλού. Σε ό,τι αφορά η αντιμετώπιση την αντιμετώπιση των ιδεών της ρωσικής προπαγάνδας, το εσθονικό παράδειγμα από το 2007 είναι χαρακτηριστικό. Τότε η Ρωσία επετέθη κατά της Εστονίας ε, με βάση κάποιες επιθέσεις σε μνημεία που έγιναν η αντεπίθεση, η αντιπροπαγάνδα δεν είναι αποτελεσματική. Η Εστονία χρησιμοποίησε διαφορετική μέθοδο. Προ, προτίμησε να αγνοήσει τα προπαγανδιστικά μηνύματα της Ρωσίας. Αλλά αντίθετα υπέβαλε τη δική της ρητορία που ήταν πολύ ελκυστική και αυτό το εστονικό αφήγημα ήταν πολύ πετυχημένο και δείχνει πώς θα πρέπει να σκεφτούμε και εμείς πώς θα διατυπώσουμε τη δική μας ιστορία, τη δική μας αφήγηση με μηνύματα που θα έχουν απήχηση και στους δικούς μας πληθυσμούς αλλά και στους λαούς άλλων χωρών. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρεσβευτά, αλλά και άλλοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, θα τους το δώσω. Και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω τι γίνεται με την μαζική προπαγάνδα που ξεκίνησε μετά την κατάρριψη του MH17 τις ε, πτήσεις του Μαλαισιανού αεροσκάφους. Πολύ, είναι, πολύ σημαντικές είναι τέτοιου είδους ε, δραστηριότητες. Ε, είχαμε και πριν από πέντε χρόνια την κατάρριψη αεροσκάφου στο Μολέσκ, την καταστροφή του στο Μολέσκ και τότε η ρωσική προπαγάνδα ισχυρίστηκε ότι η Πολωνία έστειλε στρατιωτικό προσωπικό που ενεπλάκη και ουσιαστικά κατηγόρησε τον ίδιο τον Πολωνό πρόεδρο για κάτι τέτοιο. Αμέσως δηλαδή ξεκίνησε την προπαγάνδα της ε, η Ρωσία που είχε ολέθρια αποτελέσματα. Ελπίζω το κέντρο σας να παρακολουθεί εκ του ε, την ε, υπόθεση και τη διαλέφραση του MH17 και την ε, συναφή προπαγάνδα της Ρωσίας. Ο κύριος Τρογεύσκη. Έχω πολύ σύντομε ερωτήσει, κύριε Πρέσβη. Ποιο είναι ο προπολογισμό σα, ποιε είναι οι δημοσιονομικέ σα προβλέψει για το μέλλον. Ευχαριστώ. Ο κύριο Κρασνοντέμσκι. Κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ένα ακόμη θέμα. Μπορεί να μην εμπίπτει στι αρμοδιότητε του κέντρου αριστεία σα, αλλά καλό θα ήταν να το λάβουμε υπόψη. Αυτή η ενισχυμένη σήμερα ρωσική προπαγάνδα και κυρίω των μέσων μαζική ενημέρωση τη Ρωσία. Ε, πέφτει σε πρόσφορο έδαφο, σε γόνιμο έδαφος, ακριβώς γιατί στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ακαδημαϊκό πρόβλημα. Έχουμε πολλές, πολλά Ινστιτούτα που ασχολούνται με τη Ρωσία, έχουμε κάποιε κατευθύνσει σπουδών πανεπιστημιακά προγράμματα που για χρόνια ολόκληρα πρόβαλαν μια εικόνα της Ρωσίας που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Και από επιστημονική άποψη είναι δυσάρεστο κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι και το κέντρο αριστείας σας έχει συνεργασία με διάφορα κέντρα και Ινστιτούτα. Και Βέβαια, εν μέρει είναι και δική μας ε, αποστολή, πολιτικό καθήκον, αλλά ίσως θα πρέπει ε, να αφυπνίσουμε και τον ακαδημαϊκό κόσμο για να θετήσει μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση και στις έρευνες ε, και στις πανεπιστημιακές σπουδές να ασχοληθεί πιο ρεαλιστικά με τη Ρωσία και να συμπεριλάβει κάποιες στρατιωτικές πτυχές στην ανάλυση. Δεν ξέρω αν έχετε συνεργασία με ευρωπαϊκά Ινστιτούτα ή με ποια τέτοια Ινστιτούτα θα έχετε στο μέλλον συνεργασία στο κέντρο αριστείας σας. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται ο κατάλογο των ομιλητών και θα δώσω το λόγο στον πρέσβη για τι απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Όντω το περιστατικό με το MH17, το αεροπλάνο που έπεσε ήταν τραγικό. Και είδαμε ότι μέσα σε μία ώρα διάφορα ρωσικά, δηλαδή διάφορα τηλεοπτική σταθμή της Ρωσίας παρουσίαζαν διαφορετικές εκδοχές των λόγων του, της ε, συντριβής με όλο και περισσότερη φαντασία και δημιουργικότητα. Γιατί? Διότι στόχος τους ήταν να αποτρέψουν από την κατά βάση αυθεντική ανάλυση των, του περιστατικού την κοινή γνώμη και κυρίως στις άλλες χώρες, δηλαδή να ε, στρέψουν την προσοχή της κοινή γνώμης σε κάτι άλλο από την πραγματικότητα της συντριβή. Ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα λοιπόν α, παραπληροφόρησης της κοινή γνώμης. Από την κοινή γνώμη και αναπτύχθηκε σε πάρα πολύ στο χρονικό διάστημα ο προπολογισμό του κέντρου μα. Χωρί σε δύο τμήματα έχουμε το λειτουργικό, τον επιχειρησιακό προπολογισμό που μας επιτρέπει να λειτουργούμε και καλύπτεται πλήρως από τη λετωνική κυβέρνηση και ο, το κοινό, τον πιο σημαντικό προπολογισμό μας που καλύπτει την διεξαγωγή διαφορών επιχειρήσεων και έργων. Έχουμε συνολικά 3 εκατομμύρια ευρώ στη διάθεσή μας το μέγιστο μέρος των οποίων καλύπτει η λετωνική κυβέρνηση. Έχουμε για την επιχειρησιακή δουλειά 500.000 ευρώ και έχουμε και ορισμένε ε, θελοντικές συνεισφορές στη χρηματοδότησή μας. Στη συνεργασία τώρα με άλλα όργανα. Είναι καινούριο το κέντρο μας. Μόλις ένα χρόνο τώρα έχουμε που ξεκινήσαμε ως ε, διεθνέ Θεσμικό Όργανο, διεθνή θεσμό. Από την 1η Σεπτεμβρίου του 2014 έχουμε την υπαγωγή και τη σχέση με τον ΝΑΤΟ. Έχουμε επαφέ με διάφορα ακαδημαϊκά ερευνητικά κέντρα της Λετωνίας, αλλά και άλλα. Πανεπιστημιακά, πανεπιστημιακούς φορείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γερμανία όλο και περισσότερο δηλαδή ανοίγουμε το πεδίο των ενδιαφερόντων μας αναπτύσσοντας παράλληλα τις προοπτικές μας. Έχουμε ξεκινήσει συνεργασία με πολωνικά, εσθονικά πανεπιστήμια, ε, το στο Τάρτο και συνεχίζουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ τον πρέσβη για την άκρος ενδιαφέρουσα αυτή τοποθέτηση για την υποεπιτροπή μας θα θέλαμε πάρα πολύ να μπορούσατε να μείνετε και να μας ενημερώσετε κι άλλο για την πρόοδο των επιχειρήσεων ε, του κέντρου υπεροχής. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Παρακαλώ αγαπητοί συναλφοί, μείνετε στην αίθουσα, διότι ξεκινούμε αμέσως τη δημόσια κρόαση για την ε, αναθεώρηση της συνθήκης περί μη διάδοσης των πυρηνικών. Ευχαριστώ ιδιαίτερος τον πρεσβευτή Ηλισέγεφ και τον ε, πρεσβευτή Κάκλινς για τις τοποθετήσει τοποθετήσεις τους αυτό το ενδιαφέρον θέμα της ημερήσια διάταξης. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. We start. Uh, Ξεκινάμε, προχωράμε μάλλον στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Τη δημόσια ακρόαση για την αναθεώρηση της συνθήκης ε, περί μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, NTP. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας. Θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας για κάποιες εισαγωγικές ομιλίες. Πρώτα θα ακούσουμε τον κύριο Όλιβερ Μάιερ, που είναι αναλυτής από ένα γερμανικό Ινστιτούτο. Θα μας παρουσιάσει ως πρώτος ομιλητής ε, τις απόψεις του μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρεβέκα Τζόνσον που εκπροσωπεί το Ινστιτούτο Ακρονίμιο Μέτρα το Λονδίνο ε, Ινστιτούτο που ασχολείται με τη διπλωματία του αφοπλισμού και θα ακούσουμε και έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ΕΙΕΔ, την κυρία Κλάραγκαν, που είναι τμήματάρχης της μονάδας ε, αφοπλισμού και μη διάδοσης. Είχαμε εκτενή συζητήση σήμερα το πρωί. Δεν μας έχει μείνει πολλούς χρόνος, γι' αυτό περνάμε κατευθείαν στις παρουσιάσεις των καλεσμένων μας. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο Όλιβερ Μάιερ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την πρόσκλησή του και για τη διοργάνωση του σεμιναρίου αυτού. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την πρόεδρο, για την παγκόσμια πυρηνική ε, τάξη και είναι φυσικά πολύ επίκαιρο το θέμα σε ό,τι αφορά και τις προετοιμασίες του, της διάσκεψης NPT. Σε τρεις μήνες ξεκινάει άλλωστε το συνέδριο. Και θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να, καταλήξει σε μια ενιαία θέση. Πριν από πέντε χρόνια και εγώ και η Ρεμπέκα μιλήσαμε πριν από το τελευταίο της σχετικό συνέδριο και ε, έχω τις σημειώσεις μου για αυτά που είπαμε πριν τότε. Ήταν πολύ διαφορετική το κλίμα, όπως θα θυμάστε, μετά την ομιλία του Πρόεδρου Ομπάμα για τη μηδονική χρήση και υπήρχε κάποια ελπίδα ότι θα γίνονταν ε, κάποια πρόοδος στην ε, διεθνή ασφάλεια σε ό,τι αφορά τη χρήση πυρηνικών όπλων. Σήμερα τα όπλα μαζικής καταστροφής και ιδιαίτερα τα πυρηνικά όπλα εξακολουθούν να αποτελούν απειλή για την ε, διεθνή ασφάλεια. Πιο μεγάλη ουσιαστικά απειλή σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια. Η συνθήκη NPT για τη μη διάδοση των όπλων αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της απειλή αυτής. Ωστόσο, έχει μείνει λίγη αισιοδοξία σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια πριν ε, την προηγούμενη εβδομάδα. Η σχετική εκτίμηση έχει έρθει σε επίπεδο έκτακτης ανάγκης ουσιαστικά στο πιο υψηλό επίπεδο έκτακτης ανάγκης ε, στα τελευταία 30 χρόνια και έχουν, ε, έχετε ότι έχουν σταματήσει οι προσπάθειες για τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων. Η αντίδραση, νομίζω, του κυρίου Ομπάμα για πρώτη φορά ήταν ότι στην ομιλία του για πρώτη φορά δεν αναφέρθηκε το θέμα καν των πυρηνικών όπλων. Και δεν είναι και μόνος ο πρόεδρος Ομπάμα. Κανένα από τα άλλα οκτώ κράτη δεν ε, εξετάζει σοβαρές μειώσεις ε, στα πυρηνικά όπλα ή μια αλλαγή στην πυρηνική νοοτροπία. Το βασικό λοιπόν ερώτημα που θα ήθελα να θέσω σήμερα είναι το εξή. Ποιο είναι το επίπεδο φιλοδεξία για τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη για την ενίσχυση τη πυρηνική τάξη. Αυτό το ερώτημα και η απάντησή του θα πρέπει να διέπει τις συζητήσεις σα σε ό,τι αφορά την διάσκεψη NPT που θα ξεκινήσει στα τέλη Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει και υποστηρίζει πάντα τα καθεστώτα ε, μη διάδοσης. Αλλά η έλλειψη προόδου για τον έλεγχο των πρινικών όπλων νομίζω ότι τοποθετεί επιπλέον ε, ευθύνη πάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να εργαστεί υπέρ της ε, ενίσχυσης των εργαλειών μη διάδοσης. Έξι σημεία θέλω να τονίσω. Εν συντομία, δύο για τη μη διάδοση και δύο για τι θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη πρόκληση είναι η έλλειψη δέσμευση από τα κράτη που έχουν πυρηνικά όπλα. Η κατάσταση είναι αρκετά απεσή έντοξη. Δεν έχει σημειωθεί την τρίπροδο τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι δύο μεγάλες, χώρε. Ε, χώρες, ε, η ΙΠΑ και η Ρωσία, μειώνουν τον αριθμό των πυρηνικών όπλων τους, αλλά ανανεώνουν τα οπλοστάσια τους εκ παραλλήλου. Κάθε χρόνο τα κράτη αυτά προξοδεύουν 100 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για τη διατήρηση των πυρηνικών τους όπλους. Αν και φυσικά είναι πολύ ανακριβή τα στοιχεία αυτά γιατί δεν έχουμε πληροφορίες. Όπως ξέρετε, οι χώρες, ε, οι προσυπογράφουσες του NPT πρότειναν την προηγούμενη φορά συγκεκριμένα μέτρα να εφαρμοστούν και μία αξιολόγηση των δεσμεύσεων αυτών, ιδιαίτερα των δεσμεύσεων που έγιναν το 2002 θα δεικνύουν ότι μόνο εν μέρη έχουν τηρήσει αυτά, αυτές οι δεσμεύσεις. Κάποιες από αυτές τις δεσμεύσεις ε, έχουν τηρηθεί, αλλά γενικά σε ό,τι αφορά τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων δεν τηρήθηκαν οι δεσμεύσεις ε, και κάποιες αρνητικές ε, εξέλιξεις στο διεθνές προσκήνιο από το 2010 καταδεικνύουν ότι το σχέδιο δράσης δεν θα πρέπει να αποτελεί πλέον τη βάση για την ε, συζήτηση για τη μη διάδοση. Θεωρώ ότι αυτό το επιχείρημα είναι επικίνδυνο. Αυτό αγνοεί το σχέδιο δράσης τότε. Ουσιαστικά περιέγραφε το status quo και θα αποτελούσε ένα πάρα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο αν ε, τα κράτη ουσιαστικά θεωρούσαν ότι μπορούν να ερμηνεύουν τις δεσμεύσεις τους ανάλογα με το διεθνές προσκήνιο. Δεύτερο στοιχείο, η επάνωδος των πυρηνικών όπλων, ιδιαίτερα στην Ασία, αλλά και για την Ευρώπη. Πολλοί πολιτικοί θύνοντες ε, ε, παρακολουθούν την ε, επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία που ασκεί μεγάλη πίεση στην συμφωνία NPT γιατί έχουν ε, παραβιαστεί οι εγγυήσει ε, που δόθηκαν στο Μνημόνιο Συμφωνίας ε, που θεωρούν ότι τα κράτη-μέλη για τη... που δεν έχουν πυρηνικά όπλα δεσμεύονται να μην ακολουθήσουν τέτοια προγράμματα. Η Ρωσία, η ΙΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να κοιτάξουμε κατά πόσον θα θεωρηθούν ένοχες από τις άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις τους. Για να μην γίνει λοιπόν αυτό, τα πυρηνικά κράτη και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενισχύσουν και να καταστήσουν πιο δεσμευτικές τις εγγύησεις ασφαλείας. Ευγενικά, η πρόεδρος παρακαλεί τον ομιλητή να μιλάει πιο αργά. Σε άλλους τομείς όπου έχουμε πρόοδο για την πυρηνικό αφοπλισμό είναι η συζήτηση για την ε, ανθρωπιστική ανθρωπιστικό αντίκτυο. Η Ρεμπέκα θα το συζητήσει αυτό, άρα δεν πρόκειται να επεκταθώ ιδιαίτερω. Να πω μόνο ότι πρόκειται για έναν τομέα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική και εκθετική εξέλιξη που έχει ανανεώσει τη συζήτηση για τον αφοπλισμό. Σε πολλές χώρες όπως και στη Γερμανία η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να σημειώσει μια μετάβαση της όλης συζήτησης σε άλλους τομείς. Βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να φροντίσουμε ότι οι προσπάθειες για από να μεμοποιηθούν τα πρινικά έργα, τα πυρηνικά όπλα, δεν θα πρέπει να αποδυναμωθούν. Τώρα, για τη μη διάδοση. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τις χώρες που δεν ε, συμμορφώνονται. Η Βόρειος Κορέα, το Ιράν. Για τη Βόρειο Κορέα νομίζω ότι το, η επίλυση θα είναι απίθανη έως αδύνατη. Όσο θεωρούνται τα πυρηνικά όπλα, η απότερη και η μεγαλύτερη εγγύηση κατά της εισβολής των ΙΠΑ. Σε ό,τι αφορά τον ε, Ιρά, το Ιράν, υπάρχουν, ε, έχουν ξεπεραστεί οι βασικές και θεμελιώτες διαφορές ε, για τα θέματα αυτά και η συμφωνία για ένα σχέδιο δράσης θα, υπήξε, θα έδινε μια μεγάλη όθηση στο NPT. Και αυτό που θα βελτίωνε τις πιθανότητες επιτυχίες επειδή το Ιράν θα συνεχίσει να έχει την προεδρία των ε, κινήματος των αδεσμεύτων. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχε νόημα να προσπαθήσουμε να μεταφράσουμε την πρόοδο που έχουμε δει στι συνομιλίε ε, με το Ιράν σε συγκεκριμένε δεσμεύσει, ιδιαίτερα για εργαλεία μη δέσμευση. Κάποιε εγγυήσει, δηλαδή και ιδιαίτερα την ικανότητα τη IAA να ε, ερευνήσει τι αρχιωτικές πτυχέ των πυρηνικών προγραμμάτων και μπορούμε να κοιτάξουμε στι ερεταπαντήσει πιο πολλέ λεπτομέρειε. Έχω συμπεριλάβει και στο φάκελό σα πιο πολλέ λεπτομέρειε. Η ηρωνία είναι ότι ενώ υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα να ενισχυθούν τα εργαλεία μη διάδοση σε σχέση με πριν από πέντε χρόνια, εξακολουθεί να είναι δύσκολο να υπάρξουν αυτά τα ωφέλη όσο δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει πρόοδος στον πυρηνικό αφοπλισμό. Γιατί εξακολουθούν να μην υπάρχει ουσιαστική πρόοδο σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό. Δύο σύντομε παρατηρήσει για, το πώς, για τον δυνατό ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βράχει πρόθεσμα. Νομίζω ότι η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να συμφωνήσει σε μια μελλοντοστραφή, αν θέλετε, ε, κοινή θέση. Και το βασικό ερώτημα και πάλι που ανακύπτει είναι τι επίπεδο φιλοδοξία πρέπει να επιδιώξουν τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει μια απάντηση στο ερώτημα αυτό στι διαπραγματεύσει για μια τέτοια απόφαση. Και κατά το παρελθόν, οι συζητήσει αυτέ για τι κοινέ θέσει ήταν σπάνιε περιστάσει όπου τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκαστικά ε, έπρεπε να συμφωνήσουν για το πώς θέλουν να περιορίσουν το μέλλον των πρινικών όπλων. Τα κράτη-μέλη θεωρώ ότι θα πρέπει να βρουν κοινό τόπο αυτή τη φορά. Ωστόσο, η συμφωνία σε μια κοινή θέση δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Ο πρινικός αφοπλισμός ε, έχει λάβει γενικά πολύ λιγότερη προσοχή στο παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σπάνιες περιπτώσεις έχει ξεπεράσει τον ε, χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Και σε μέσα γραμμές αυτό δεν περιλαμβάνει αυτά που θέλουν να αποδεχτούν τα μη πυρηνικά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν επαρκεί λοιπόν αυτή η προσέγγιση που είχαμε ως τώρα για τον πυρηνικό αφοπλισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σημειώσει καλύτερα αποτελέσματα φέτος να σκεφτεί και το σημαντικό ρόλο τη συζήτηση του ανθρωπιστικού αντικτύπου. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι δυνατόν, γιατί για πρώτη φορά όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με την εξαίρεση τη Γαλλία, συμμετείχαν στην ε, συνεδρίαση τη Βιέννη το Δεκέμβριο. Η μακροπρόθεσμη πρόκληση θα είναι να βρεθεί ένα σχέδιο μη διάδοση και αφοπλισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των συζητήσεων για μια αναθεωρημένη ε, στρατηγική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει αυτή τη μεταρρύθμιση η οποία έπρεπε να έχει γίνει πριν από καιρό. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το 2003 οι προσπάθειες για την ε, στρατηγική ασφαλεία και κατά τον ε, όπλο μαζικής καταστροφής προκλήθηκαν ε, ουσιαστικά από δύο περιστατικά από την 10η Σεπτεμβρίου και τον πόλεμο στο Ιράκ η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και η νέα τέτοια στρατηγική του WNB θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτά τα γεγονότα για να κλείσουν κάποια από τα χάσματα που υπάρχουν στην σχετική πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ρεπίκα Τζόνσον. Χωρίς μικρόφωνο. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκλήθη να εξετάσω την κατάσταση πιθανές εξελίξεις και μόλις τώρα και να κόψω πέντε λεπτά από το αρχικό μου κείμενο. Με ακούτε καλά? Όχι. Θα προσπαθήσω λοιπόν πάρα πολύ σύντομα να εκθέσω τις ε, τέσσερις κύριες προκλήσεις. Την πρώτη ήδη την ε, αναέπηξε ο Όλιβερ η απουσία δηλαδή εφαρμογής όχι μόνο των συμφωνιών για τον εφοπλισμό του 2010 που ήταν συνενετικές αλλά και του μακροπρόθεσμου ζητήματος για την υλοποίηση που ανάγεται στην πρώτη διάσκεψη κιόλα της συμφωνίας για τη μη διάθεση μετά τη θέση της εφαρμογή του 1970 όπου τότε είχαν ιδιαίτερα επικεντρωθεί στην απαγόρευση των δοκιμών και αργότερα μια σταδιακή διαδικασία που είχε συνενετικά προχωρήσει το 2000 από τα πυρηνικά κράτη. Κύριες προκλήσεις λοιπόν εντοπίζονται στη Μέση Ανατολή. Και πάλι περιορισμένος ο χρόνος μου και οι διάφορες συνθήκες που αντιμετωπίσω δεν δεν μου επιτρέπουν να εκθέσω πιο διεξοδικά τα ζητήματα τα σχετικά με την ε, διάσκεψη 2012. Έγινε μια προσπάθεια για ανάπτυξη αυτής της ε, ε, διάσκεψης με την υποστήριξη δεύτερα της Φιλανδίας ε, αλλά και οι πολιτικές και λοιπές ε, συνθήκες δεν επιτρέπουν κυρίως η παρουσία των πυρηνικών στο Ισραήλ και θέματα που έχουν να κάνουν με τα χημικά της Συρίας τα όπλα μαζικής καταστροφής, όλα αυτά τα ζητήματα που ήθελε να εξετάσει. Είναι ζητήματα λοιπόν τα οποία θα είναι δύσκολο να καλύψει η διάσκεψη 2015 για τη συνθήκη περιμηδιάδοσης. Ε, ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τη διάδοση και εδώ εντάσσω και την πυρηνική ασφάλεια που δεν ήταν αρχικά ζήτημα της μη διάδοσης αλλά μετά την ε, επίθεση της 11 Σεπτεμβρίου μπήκε στο θεματολόγιο και με πρωτοβουλία του Πρόεδρου Μπούς και με τις διασκέψεις για τα πυρηνικά του Πρόεδρου Ομπάμα με μια προοπτική δυτική κυρίως και τώρα και έτσι κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες εμπλέκονται και συμμετέχουν σε αυτές τις διασκέψεις για την πυρηνική ασφάλεια με τη δυσφορία παρόλα αυτά που υπάρχει και ανέφερε και ο Λιβέρ τα θέματα τα σχετικά με το Ιράν ε, και δεν θα πω στις λεπτομέρειες και το τέταρτο, ε, ο προκλήσεων για μετά το 2015 που θα ήθελα να υπογραμμίσω κυρίως τις προοπτικές που είχαμε εντοπίσει το 2010 που γινόταν λόγος κυρίως για την πυρηνική αναγέννηση και μετά το φούτι βέβαια και το τσουνάμι προκάλεσε την καταστροφή εκεί. Αυτό που θέλουμε ιδιαίτερα εδώ είναι ε, να ρίξουμε κάπως τους τόνους σε σχέση με την πυρηνική αναγέννηση πριν την πυρηνική καταστροφή της Φουκοσίμα, αλλά μια ε, προσέγγιση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιορισμένη κλίμακα και εύρου χρήση, σε ιατρικέ κυρίω ε, έρευνε και καινοτομία της πυρηνικής ενέργειας, αλλά πάντως όχι την εκτεταμένη αυτή ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και κυρίως ανησυχίες σε σχέση με την ασφάλεια. Και θα επικεντρωθώ τώρα στι λοιπέ μου παρατηρήσει στα κύρια ζητήματα του πυρηνικού αφοπλισμού. Πάλι μέσω του, του ιστορικού υποβάθρου, το οποίο ασφαλώ γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θα ξεκινήσω λοιπόν με το άρθρο 6, το οποίο ρητά ενσωματώνει τις υποχρεώσεις για πυρηνικό αφοπλισμό όχι μόνο των πυρηνικών δυνάμεων αλλά όλων των κρατών ως ευθύνη τους για την εξασφάλιση των συνθήκων, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στο να συζητούμε γιατί ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες οι οποίες προχώρησαν από το 2010 έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω το άρθρο 7 που δεν ακούγεται πολύ συχνά σε σχέση με τον αφοπλισμό, αλλά μιλά για μια ελεύθερη ζώνη πυρηνικών που πάλι υποστηρίζουν όλα τα κράτη. Η συμφωνία λοιπόν του 1996, η Σφαιρική Συμφωνία για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών ε, ε, ορίζει τα στοιχεία σχετικά με τον πυρηνικό αφοπλισμό και έχουμε να κάνουμε με, τα πυρηνικά, με τις πυρηνικές δυνάμεις που πρόκειται να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία για την απαγόρευση των ε, πυρηνικών δοκιμών. Προχώρησε αυτή η εξέλιξη στο 1995 με διαπραγματεύσεις που ε, ακολούθησαν την αποτυχία της ε, διάσκεψης του 1994 και που θα οδηγούσαν σε μία απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών με πίεση ώστε η διάσκεψη του 1995 που παρέτεινε την ε, σύμβαση περί μη διάδοσης, ύστερα από 25 χρόνια λειτουργίας της, χαρακτηρίστηκε ως επιτυχής. Και αυτή νομίζω ήταν μια πολύ σημαντική πτυχή με συγχωρείτε, ξαναψάχνω λίγο τις ε, διαφάνειε στον υπολογιστή μου. 95, λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 1995, όπου ορίζονται αρχές και ε, στόχοι με ουσιαστικά και αποτελεσματικά βήματα για τον πυρηνικό αφοπλισμό και την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών που μεταφράζονται σε, μια σε χίλιες περίπου ε, διασκέψεις αναθεώρησης με 30 περίπου βήματα αναθεώρησης μονομερή, διμερή, πολυμερή βήματα και με λύπη μου πρέπει να πω ότι το πρόγραμμα δράση του 2010 οπισθοδρομεί σε σχέση με αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί το 2000 διότι δεν υλοποιήθηκαν αυτές οι δεσμεύσεις και έτσι πάμε τώρα με προοπτική το 2015 όπου απέχουμε όχι μόνο από την υλοποίηση των 13 εκείνων βημάτων του 2000 αλλά και από τις δεσμεύσεις του 2010. Ούτε αυτές έχουν υλοποιηθεί. Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Εν γέννη, οι πυρηνικές δυνάμεις ε, επικεντρώνουν την προσοχή τη δράση 4 και 5 που δεν έχουν υλοποιήσει πάλι, αλλά σε αυτές επικεντρώνεται περιορισμός δηλαδή, των δυνάμεων, των μονάδων, των κινδύνων. Με στόχο τη μείωση του κινδύνου γενικότερα. Αλλά εγώ θα ήθελα να στραφώ σε δύο άλλα ζητήματα. Τη δράση παριθμών 3 καταρχάς η οποία με στεναρό τρόπο αντυχεί το κεντρικό μήνυμα των 13 βημάτων της Συμφωνίας του 2000 που ήταν η ανεπιφύλακτη δέσμευση για ολοκλήρωση από τις πυρηνικές δυνάμεις της καταστροφής του πυρηνικού τους ε, δυναμικού, ξεκάθαρη δέσμευση, αλλά και το θεματολόγιο του Ομπάμα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά. Δηλαδή ανάληψη δεσμεύσεων για τη μείωση και καταστροφή κάθε τύπου πυρηνικών, ανεπτυγμένων και μη ανεπτυγμένων όπλων, μέσω, επαναλαμβάνω, μονομερών, διμερών, περιφερειακών και πολυμερών μέτρων. Θέλω επίσης να πιστήσω την προσοχή σας. Δεδομένη της πολύ δύσκολης κατάστασης το 2010, κυρίως όσον αφορά την Μέση Ανατολή, και την ε, επανεισαγωγή των 2.000 ε, μέτρων στην ε, πρόταση δράσης του 2010 και θέλω να πω ότι ήταν και ευρωπαϊκά κράτη όπως η Αυστρία, η Ιρλανδία ευτυχώς και δεν θυμάμαι πια, και άλλα κράτη, οπωσδήποτε η Αυστρία, η Ιρλανδία, τα νέα κρατημέλη με την Σουηδία ασφαλώς και την Ορβηγία που δεν ανοίξει την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πάντως είναι Ευρωπαίος εταίρος. Προσπάθησαν λοιπόν τα κράτη αυτά το ζήτημα της χρήσης των πυρηνικών όπλων που κανονικά δεν συζητείται στο πλαίσιο της ε, σύμβασης περί μη και των συνεπειών που έχουν να κάνουν με το ανθρωπιστικό διεθνές δίκαιο, απαγόρευση των ε, όπλων διασποράς, των ναρκών κατά προσωπικού και ούτω καθεξής. Να βάλουν λοιπόν αυτή την προοπτική μέσα στο θεματολόγιο για τη μη διάδοση και ξέρετε αυτό συνενετικά υιοθετήθηκε ώστε να πλαισιωθεί χωρίς να είναι θέμα ακριβώς δράσης αλλά πλαισίωση όλων των σημείων για δράση ως προς τους πυρηνικούς αφοπλισμούς γιατί επισημενόνταν και οι ανθρωπιστικές συνέπειες ιασδήποτε χρήσης πυρηνικών όπλων και η υποχρέωση για συμμόρφωση με το ισχύον διεθνές αλλά και, ε, και ε, Ε, κρατικό δίκαιο. Όλα αυτά με τις διασκέψεις που είχαμε μέχρι και τη Βιέννη, με έμφαση ιδιαίτερα όπως είπα στις ανθρωπιστικές συνέπειες. Και έτσι, με τη διάσκεψη της Βιέννης, που θα ήθελα λίγο περισσότερο να εκθέσω το συσχετισμό της για να φτάσω σε συστάσεις και προτάσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανθρωπιστική πρωτοβουλία ήταν ένα πρώτο βήμα μέσα στην ε, Σύμβαση για τη Μη Ξεκίνησε από την Ελβετία, μετά ακολούθησαν η Νέα Ζηλανδία, η Νότιο Αφρική. 150 εν όλο ήταν τα κράτη που ακολούθησαν ως μέλη της Σύμβασης περί Μη για την υπογραφή δεσμεύσεων για τις ανθρωπιστικές συνέπειες και η πρόταση από την Επιτροπή Μπλίξ που είχε ξεκινήσει η Σουηδία για την απαγόρευση κάθε τύπου πυρηνικών όπλων και στη Βιέννη είχαμε μια αναπάντηχη εξέλιξη με 157 κράτη μαζί με τον ε, Διεθνή Ερθρό Σταυρό και άλλες ανθρωπιστικές διεθνείς οργανώσεις που καταλήγουν σε συμφωνία και διαπιστώσεις αναφερόμενες ιδιαίτερα στις συνέπειες της πιθανής χρήσης ή δράσης που θα είναι καταστροφικές, μη ελεγχόμενες από εθνικά σύνορα και ω εκ τούτου συνιστά ευθύνη κάθε κράτους μέλους των συμβαλωμένων στην ε, Σύμβαση Περιμηδιάδος αλλά και οποιοδήποτε συμβαλωμένου στο Χάρτη των Εθνών με κινδύνους ε, τεράστιους για τον άνθρωπο ε, κινδύνους που δεν είχε περιγράψει προηγουμένως εθνική Συνθήκη. Όλες λοιπόν, όλα τα συμβαλώμενα μέρη και τα κράτη Αναλαμβάνω αυτή τη διάσμευση εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι συναδελφοί σας βέβαια στα Εθνικά Κοινοβούλια και στη Διακοινοβουλευτική Ένωση ε, διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα κοινοβουλευτικά όργανα και βέβαια μέσα στη συνθήκη για τη μη διάδοση παρακαλώ ε, αναπτύξτε δραστηριότητα, εξηγήστε στις κυβερνήσεις σας τι σημαίνει ακριβώς αυτή η δέσμευση της ε, Βιέννης όπως ονομάστηκε και οθήστε τους να την προωθήσουν. Μην γίνεται λόγος για ένα γενικό ψήφισμα για την ε, συνθήκη περί διάδοσης. Παρακαλώ πιέστε όσο γίνεται να προχωρήσει. Γίνεται λόγος. Ναι, αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώνετε. Καλά, σταματάω εδώ λοιπόν και πολύ ευχαρίστως να τοποθετηθώ όταν διατυπωθούν ερωτήσεις σχετικές με οποιαδήποτε πτυχή και για τη δέσμευση της ε, Βιέννης, την αυστηριακή δέσμευση, αλλά και για άλλα ζητήματα. ευχαριστώ και στο συγγνώμη που σας ε, διέκοψε, λέει η Πρόεδρος. Θα προτιμούσα να ακούσω πιο αμερόληπτες τοποθετήσεις από τους ειδικού στις δεσμεύσεις τους. Thank you very much. Uh, σας ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία που δώσατε να έρθω και να σας παρουσιάσω τις ευρωπαϊκές απόψεις και τις ευρωπαϊκές δράσεις ε, για την αποπυρηνικοποίηση. Θα επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες μας ανάψη τη επικείμενη διάσκεψη για την ιδιάδα των πυρηνικών που είναι το σημαντικότερο φετινό παγκόσμιο γεγονό για την αποπυρηνικοποίηση. Η διάσκεψη αναθεώρηση θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και προκλητική. Μικτές, ε, ανάμεικτε προοπτικέ. η ε, πρόοδος ε, δεν ήταν πολύ σημαντική μέχρι τώρα, αυτό είναι το αρνητικό και το θετικό είναι ότι το Ιράν και παράταση των, ε, των διαπραγματεύσεων ε, μέχρι τον Ιούνιο. Τώρα, ανάλογα με την πιθανή, πιθανή έκβαση ε, είναι να μην γίνει η διάσκεψη γιατί να μην είναι μια ζώνη χωρίς πυρηνικά στη Μέση Ανατολή. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα στην αξιολόγηση της προόδου της αποπυρηνικοποίησης. Το ανέφερε και η δόκτωρα Τζόνσον ε, για τον ανθρωπιστικό αντίκτυπο των πυρηνικών όπλων. Εκεί έχουμε δύο πλευρές, δύο στρατόπεδα. Η μία ε, αναφέρεται στην ε, απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών και η άλλη αφορά μια σταδιακή προοδεστική μείωση και όχι ολοσχερή, όπως η πρώτη πλευρά, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και το DPRK στη Συρία ε, δημιουργεί προβλήματα σοβαρά και ανησυχίες ό,τι αφορά τη μη διάδοση των πυρηνικών. Ε, και μία επιφύλαξη αυτή τη στιγμή. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακόμη αποκρισταλωθεί εν ώψη της διάσκεψης της θεώρησης της συνθήκης μη διάδοσης. Συνεχίζονται ε, οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωση της θέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως ε, θα ήθελα να δηλώσω το προφανές ότι θέλουμε να προασπίσουμε και να διαφυλάξουμε τη συνθήκη αυτή που είναι ακρογωνία λήθος του συστήματος αποπυρηνικοποίησης. Αυτή είναι η βασική μας προτεραιότητα. Θεωρούμε ότι η συνθήκη περί μη διάδοσης των πυρηνικών ε, είναι η ραχοκοκαλιά του παγκόσμιου συστήματος για την ε, μη διάδοση των πυρηνικών. Και με βάση το άρθρο 6 του MPT ε, έχουμε σημαντικά στοιχεία για τη μελλοντική αποπυρηνικοποίηση αλλά και χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς. Είμαστε υπέρ της οικουμενικοποίησης της συνθήκης και της έμπρακτης εφαρμογής της. Θέλουμε να συμβάλλουμε όλοι για να παραμείνει ζωντανή η ζωτική αυτή συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Θα πρέπει να εφαρμοστούν και οι τρει πυλώνε της και περιμένουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέρη να δραστηριοποιηθούν στις συζητήσεις και για τους τρεις πυλώνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δεσμευθεί να συνεργαστεί με όλα τα κράτη για αίσια έκβαση με σημαντικά αποτελέσματα της ε, διάσκεψης για την αναθεώρηση προκειμένου να χαράξουμε το δρόμο μέχρι το 2020 τότε που η NPT θα, έχει την, θα γιορτάσει την 50η επέτειο. Θέλουμε να ενισχύσουμε το παγκόσμιο καθεστώς μη ε, διάδοση των πυρηνικών προωθώντας ε, μια ισορροπημένη και θετική έκβαση της επόμενης διάσκεψης αναθεώρησης. Και θέλουμε χειροπιαστή και ρεαλιστική πρόοδο για την υλοποίηση των στόχων που αναφέρονται στην συνθήκη περιμή διάδοση. βασικό μα στόχο είναι να δημιουργήσουμε προποθέσει για ένα κόσμο χωρί πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με, τις, ε, με του στόχου και του NPT, προωθώντα την παγκόσμια σταθερότητα ε, και την παγκόσμια προσπάθεια ενόψη αυτή τη υλοποίηση του στόχου. Θέλουμε γι' αυτό μία περιεκτική, ισορροπημένη και έμπρακτη εφαρμογή του σχεδίου δράσης ε, της διάσκεψης αναθεώρησης που ήταν ο κοινό οδικό χάρτη εν ώψη τη επόμενη διάσκεψη. Επίση, ζητούμε από όλα τα συμβαλόμενα μέρη τη συνθήκη ε, να εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο δράση. Όπω ε, είπαμε και προηγουμένω, δύο πιθανά σημαντικά θέματα τη διάσκεψη αναθεώρηση είναι η άλλη διάσκεψη για τα όπλα μαζικής καταστροφής και μία σχετικά ελεύθερη ζώνη για τα όπλα αυτά στη Μέση Ανατολή και επίσης μία συζήτηση για τις ανθρωπιστικές συνέπειες των πυρηνικών όπλων. Βέβαια πολλές άλλες διασκέψεις θα διεξαχθούν παράλληλα όπως είχαμε στο Όσλο το 2013, στο Νάιρετ και στη Βιέννη το 2014. Ξέρω ότι ο χρόνος μας πιέζει κυρία Πρόεδρε. Έχω και άλλες ε, πληροφορίες ως προς τις λεπτομέρειες, αλλά προτιμώ να σταματήσω εδώ για να ακούσουμε τις ερωτήσεις των συναδέλφων. Μάλιστα. Μπορείτε να επεκταθείτε περισσότερο στα θέματα αυτά κατά τις απαντήσεις που θα δώσετε. Η κυρία Σαμπάιος. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά Γι' αυτό σας παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη μου χαρά και τη διεξαγωγή αυτής της δημόσιας ακρόασης. Είναι πολύ σημαντική αυτή η δημόσια ακρόαση για τα μέλη της υποεπιτροπής μας, γιατί θέλουμε να ζούμε σε έναν κόσμο ασφαλή και σε ένα προστατευμένο περιβάλλον και από αυτή την άποψη η κατάργηση των πυρηνικών είναι σημαντικό στοιχείο μιας τέτοιας ασφάλειας και θα ήθελα να στεφτεί με επιτυχία η επόμενη διάσκεψη αναθεώρησης ε, της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Δεδομένου όμως των τελευταίων εξελίξεων, ιδιαίτερα στην Ουκρανία, αλλά όχι μόνο, ε, και σε διάφορες άλλες περιοχές που δεν λειτουργήσαν αυτά τα εχέγγυα ασφάλεια, διαρωτώμαστε αν είναι όντως προοπτικές για τη διάσκεψη αυτή. Θα βελτιωθεί η συνθήκη περί μη διάδοση των πυρηνικών ή μήπως θα επιδεινωθεί. Εμένα με απασχολούν ιδιαίτερα οι ανθρωπιστικές συνέπειες της κατάστασης. Γιατί αυτή κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα των χωρών. Γιατί οι ανθρωπιστικές συνέπειες είναι μιζο ζήτημα και το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας το ίδιο. Το ανέφερε ο κύριος Μάγερ στη δική του παρουσίαση. Δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουν ε, τα πυρηνικά όπλα, σε ποια χέρια θα καταλήξουν. Και δεν ξέρουμε αν κάποια στιγμή ένα κράτος που διαθέτει πυρηνικά όπλα θα διστάσει να τα χρησιμοποιήσει βάρος των ίδιων των πολιτών του. Το θέμα λοιπόν το ανθρωπιστικό είναι ένα σημαντικό θέμα και το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας άλλο εξίσου σημαντικό. Θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη της συνθήκης να, να εξετάσουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη διάσκεψη αναθεώρησης του 2015. και τους λίγους μήνες που μας χωρίζουν από τη διάσκεψη θα μπορούσαν οι χώρες μέλη να ασχοληθούν με όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να ασχοληθούμε και με την ανθρωπιστική διάσταση αλλά και με την πυρηνική ασφάλεια. Τι θα γίνει αν αυτή η πυρηνική τεχνολογία πέσει σε χέρια κακοποιών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπώνησε σχετικό ψήφισμα και η Δόκτωρ Τζόνσον μας ε, είπε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς ως πολιτικοί. Είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφανθεί με ενιαία φωνή ε, στο θέμα αυτό για να ασκήσει επιρροή στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να διατρανώσουμε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις προσδοκίες μας από την επικείμενη διάσκεψη αναθεώρησης τις συνθήκες για τη μη των πυρηνικών. Είμαστε λοιπόν ευρωβουλευτές και ταυτόχρονα πολιτικοί ηθήνοντες ε, που έχουμε σχέση φυσικά και με την εσωτερική πολιτική των χωρών μας. Ε, γι' αυτό και θα πρέπει να ασκήσουμε την επιρροή μας ε, και στην εσωτερική μας πολιτική. Η πατρίδα μου η Σουηδία ασχολείται με τα θέματα πυρηνικού αφοπλισμού και θα πρέπει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποκρισταλώσουμε τη θέση μας και να την μεταφέρουμε και στις πατρίδες μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θέρμα τους καλεσμένους και να σας ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση γιατί ήμουν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Μεταφορών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τζόνσον και την κυρία Γκάνσλαντ για τις ε, ομιλίες τους και να κάνω και ένα σχόλιο. Ε, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας κυρία Πρόεδρε ότι όλοι οι καλεσμένοι μας θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδεολογία. Τα πάνελ θα πρέπει να είναι ε, πολύμορφα, πλουραλιστικά και να πηχούν ένα ευρύ φάσμα ιδεών. και εμείς στην υποεπιτροπή μας δεν έχουμε μία απόλυτη σύμπνοια απόψεων και χαίρομαι για την πολυμορφία που υπάρχει. Η Δόκτωρ Τζόνσον όχι μόνο είναι εμπειρογνώμων ή δήμων, όπως φαίνεται και από τα γραπτά της, αλλά ταυτόχρονα έχει σημαντική κοινωνική δράση σε έναν τομέα που εξαιτία της αδιαφάνειας, εξαιτία της ιστορίας, αλλά και της καθημερινότητας και όλων αυτών των σημείων που μας προβληματίζουν, ε, θα πρέπει να την ακούσουμε γιατί έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται σε επικίνδυνη κατάσταση και ε, υφίστανται τις συνέπειες αυτής της ύπαρξης των πυρηνικών. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω μια ερώτηση προς την κυρία Τζόνσον. Υπάρχει ένα θέμα της μη διάδοσης που αφορά την καταστροφή των πυρηνικών. Πώς θα χρηστεύσουμε θα παροπλήσουμε το πυρηνικό επλοστάσιο. Είναι αυτό το έργο ένα πολιτικό και κοινωνικό καθήκον. Δεν είναι μόνο το τέλος ε, των εργασιών. Φυσικά θα πρέπει να γίνει και μια προεργασία στην πρόληψη. Αλλά καλό θα ήταν η πρόληψη να συνοδευτεί και με μια προσπάθεια μείωσης του πυρηνικού οπλοστασίου. Πυρηνικού παροπλισμού και αφοπλισμού γιατί δεν έχει νόημα να επικεντρωνόμαστε στην πρόληψη και ταυτόχρονα το πυρηνικό ε, οπλοστάσιο να μεγεθύνεται σταδιακά. Και η κυρία Γκάτσλαντ. Θα ήθελα να ρωτήσω και εγώ, όπως και η κυρία Σεβάγιος, ε, πώς μπορεί κατά τη γνώμη σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλει στο να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα και να αποκτήσουν περισσότερη προβολή αυτά τα θέματα ώστε να καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι ο πυρηνικός αφοπλισμός. Ευχαριστώ. Mrs. Ward. Ward. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πολύ λυπάμαι που δεν ε, μπόρεσα να είμαι εδώ ε, στην αρχή της συνεδρίασης ε, και με απασχολεί πάρα πολύ το ζήτημα αυτό και πρέπει να πω ότι έκανα συνεντεύξεις και επιπλέον προσωπικό γιατί με ε, έχουν κατακλείσει τα καθήκοντά μου ε, ως Ευρωβουλευτής. Εκπροσωπώ τη Δυτική Αγγλία και το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Έχει τεράστια σημασία γιατί πολλοί στην εκλογική μου περιφέρεια έχουν βρεθεί αναγκαστικά να δουλεύουν στην πυρηνική βιομηχανία, το οποίο αυτό που θα ήθελα να κάνουν είναι να έχουν μια αξιοπρεπή δουλειά που να τους δίνει μια ασφαλή ζωή. Δεν είναι πολύ ασφαλές λοιπόν για μια πόλη όταν είναι μια πόλη που εξαρτάται από τη μηχανή αυτή. Αυτά εισαγωγικά και το θέμα λοιπόν αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα γιατί εκπροσωπώ άτομα τα οποία βλέπουμε ότι η ζωή τους έχει ε, κατακλειστεί από το οικονομικό αυτό επιχείρημα. Είχα επαφέ επίση με τον Πράσινο Σταυρό και πήγα σε μια αποστολή στη Φοκουσίμα με τον Πράσινο Σταυρό στι αρχέ του έτου για να συζητήσουμε για τα πυρηνικά εργοστάσια. Τι κάνει ο Πράσινο Σταυρό, θέλει να αποχαρακτηριστούν στρατιωτικέ πυρηνικέ εγκαταστάσει μετά από το τέρμα του ψυχρού πολέμου. Ένας συνάδελφος το είπε αυτό προηγουμένως πώς θα το πετύχουμε αυτό. Υπάρχουν οργανώσεις. Ο Πράσινος Σταυρός ασχολείται με αυτό το θέμα και η εμπειρία μου από τη συνεργασία μαζί τους είναι πολύ αισιοδοξή. Γιατί αυτά τα πολύ δύσκολα καθήκοντα και επικίνδυνα καθήκοντα και σε ό,τι αφορά την πολιτική αλλά και σε ό,τι αφορά τις πρακτικές λεπτομέρειες τα αναλαμβάνουν σε ό,τι αφορά την, ε, τον αποχαρακτηρισμό, την ε, δημιουργία ασφαλών ε, τέτοιων εγκαταστάσεων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Έχω παραστεί και στο παρελθόν σε τέτοιες ε, εκδηλώσεις στο Κοινοβούλιο. Με μεγάλη μου χαρά, γιατί μου αρέσει πολύ η συνεργασία με την ε, κοινωνία των πολιτών, με τους νέους και η διάσκεψη της Βιέννης είχε μεγάλη εστίαση στους νέους. Με μεγάλη μου χαρά λοιπόν είδα ότι μπόρεσα να συμμετάσχω και εδώ. Πήγα λοιπόν και στη Βιέννη και στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών και συμμετείχα και στην Υπουργική Διάσκεψη της ε, Αυστριακής Κυβέρνησης. Στην πρώτο μου μήνα ως βουλευτής ε, προσυπέγραψα την δέσμευση ICAM και θεωρώ λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δραστηριοποιηθεί πιο έντονα το 2010 και το 2005 πριν από την αναθεώρηση της ε, διάσκεψης ε, της συμφωνίας NPT προσυπογράψαμε τέτοια ε, ψηφίσματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να περάσει ένα ψήφισμα που θα ζητάει μια συμφωνία η οποία θα απαγορεύει τα πρινικά όπλα. Μια συμφωνία στην οποία να συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη που θα προωθεί τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να θυμόμαστε γιατί υπάρχει καν η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επέτειο του Μεγάλου Πολέμου και της τεράστιας απώλειας ζώων. Δεν θα πρέπει λοιπόν να βρεθούμε σε θέση να διαδίδουμε όπλα με ακόμα πιο μεγάλη δυνατότητα καταστροφής. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με μία φωνή σε ό,τι αφορά τον πυρηνικό αφοπλισμό και τη μη διάδοση. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρο. Η κυρία Λούζινγκ τώρα έχει το λόγο. Α, όχι. Δεν ζητάει το λόγο. Παρανόηση. Ο κύριο Σαφχάζερ. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω επί τη ουσία. Με εξέπληξε η, παρέμβαση του πρέσβη της Ουκρανίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Άλλο είναι το θέμα της ημερήσιας διάταξης που εξετάζουμε τώρα, κύριε συνάδελφε. Ναι, ναι, αλλά είναι θέμα ουσίας. Γιατί ακούσαμε τον Ουκρανό χωρίς να ακούσουμε τον το Ρώσο πρέσβη. Δεύτερη φορά που προσκαλούμε τον Ουκρανό πρέσβη. Νομίζω ότι σκόπιμο θα ήταν να καλέσουμε και την άλλη πλευρά. μάλιστα απουσίαζα από, γιατί πήγα να ακούσω τον Ρώσο πρέσβη στην ε, επιτροπή που εξέτασε αυτό το θέμα της Ρωσίας. Υποτίθεται θέλουμε να είμαστε μερόληπτοι, αντικειμενικοί, ουδέτεροι και να διαμορφώσουμε τη δική μας γνώμη. Γι' αυτό και οφείλουμε να κρατούμε ίσες αποστάσεις και να καλούμε και τις δύο πλευρές αν θέλουμε πραγματικά να διαμορφώσουμε γνώμη για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Κύριε Στετίνα. Eh, Θα ήθελα να απαντήσω στον προηγούμενο μιλητή. Στον αξιότιμο βουλευτή. Εν συντομία, δεν θέλω να είμαι ουδέτερος εγώ σε αυτή τη σύγκρουση. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ακούμε τους Ρώσους πρέσβεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η Πρόεδρος, θα ήθελα να πάρω και εγώ το λόγο τώρα ως ε, μέλος της Υποεπιτροπής. Και κυρίως θα ήθελα να στραφώ προς τον κύριο Όλιβερ Μάιερ να μας ε, εξηγήσει πώς σκέφτεται και για το θέμα αυτό. Να μιλήσω προνικά. γιατί θα είναι σημαντικό να μιλάω τη μητρική μου γλώσσα. Mm. Θυμάμαι συνεχώς την ημέρα της 7ης Απριλίου του 2007 όταν υπεγράφει η Συμφωνία της Νέας Αρχής και ξεκίνησε η διαδικασία της κύρωσης. Πριν όμως ολοκληρωθεί η διαδικασία της κύρωσης Ε, μιλήσατε όλοι για το γεγονό ότι μας κατέκλυσε ένα κύμα αισιοδοξία με το πρόγραμμα του Ομπάμα. Αλλά τρεις μέρες αργότερα είχαμε την αεροπορική καταστροφή του Σμολένσκ. Και μάλιστα στις 7 Απριλίου την ίδια μέρα είχαμε και τη μεταστροφή στο Κυργιστάν, η Κυργισία οι, αργό... οι μεταγενέστερες εξελίξεις ε, σε μια περιοχή που ε, ήταν προηγουμένως ε, ζώνη σφαίρας επιρροής της Σοβιετικής Ένωσης ήταν πολύ λογικές εξελίξεις, αναμενόμενες. Ήταν εξελίξεις για τις οποίες είχαμε μιλήσει και τις οποίες είχαμε προβλέψει εδώ και πολύ καιρό. Όταν μπροστά στο, στο φως των προβολέων και με πολλή αισιοδοξία υπογράφει η Συμφωνία της Νέας Αρχής δημιουργήθηκαν πολλές ελπίδες ε, και στην δική μου πατρίδα αλλά ήδη δημιουργούνταν οι συνθήκες για την αλλαγή αυτής της κατάστασης ασφάλειας. Εγώ πραγματικά χάρηκα πολύ που άλλαξαν οι νοοτροπίες και άλλαξε και η, η άποψη των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. γιατί στο πρώτο εξάμεινο του 2007 ε, είπαν κάποιοι ότι από την που ολοκληρώθηκε η καταστροφή της Σοβιετικής Ένωσης ε, ε, ξεφορτωθήκαμε όλες τις προκλήσεις. Έχουμε τώρα την φάση της συνεργασίας. Δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε καμία άλλη πρόκληση από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ανοίγεται εποχή συνεργασίας. Τότε λοιπόν ε, γεμάτη ενθουσιασμό και αισιοδοξία υπογράφαμε τη νέα συμφωνία. Και όλα αυτά που συζητούμε σήμερα υπήρχαν στα στρατηγικά έγγραφα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Είχαμε έγγραφα που αναφερόταν στο στρατιωτικό δόγμα. Δεν αναφερόταν αμυντικό δόγμα, αλλά στρατιωτικό, πολεμικό δόγμα και την πολιτική αντίληψη της Ρωσίας ε, για την εξωτερική πολιτική τη γνωρίζαμε από τότε. Και έχω την αίσθηση ότι μετά τους ελιγμούς της Δύση και κοντά στα σύνορα της Πολωνίας και των Βαλτικών χωρών το 2009 και μετά από δηλώσεις σημαντικών πολιτικών ευθυνόντων της Ρωσίας για τη δυνατότητα χρήσης των όπλων μαζικού ολέθρου νομίζω ότι περάσαμε μια, σε μια φάση που προηγουμένως ήταν αδιανόητη, αλλά θα πρέπει να τα δούμε αυτά υπό το νέο φως και υπό, το φως αυτό που μας είπε ο πρόεδρος Κάρκλινς. Έχουμε και μια τεράστια προπαγανδιστική εκστρατεία της Ρωσίας που στηρίζεται στην ε, ε, μετάδοση του φόβου, μια εκφοβιστική προπαγανδιστική προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα να είμαι αισιόδοξη γιατί όπως και εσείς σίγουρα δεν θέλω να επικρεμάτε πάνω από το κεφάλι μας μία απειλή πυρηνικού όπλου, χρήση πυρηνικών όπλων ή όπλων μαζικής καταστροφής. Η διαδικασία όμως του πυρηνικού αφοπλισμού θα πρέπει να είναι ρεαλιστική και να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία. Πρώτα απ' όλα να λάβει υπόψη τις ουσιαστικές, τις πραγματικές απειλές δεν θα ήθελα πια να γίνουν συζητήσεις ε, που δεν θα λαμβάνουν υπόψη και τη γνώμη των δικών μας χωρών. Με την ίδια σειρά, ο κύριος Μάιερ, η κυρία Τζόνσον, κυρία, κυρία Γκάνσκαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Να προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τα σχόλια σε τρεις ομάδες δύο σύντομα και ένα πιο εκτενές. Για το θέμα της ε, ανθρωπιστικής ε, επιρροής του ανθρωπιστικού αντικτύπου και των δύο στρατοπέδων που ανέφερε. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η αντίληψη θα επικρατήσει στο νέο συνεδρίο. Η ελπίδα μου είναι οι δύο προσεγγίσεις οι οποίες σαφώς και διαφέρουν και κρύβουν μια διαφορετική φιλοσοφία, να μπορέσουν να υποστηριχθούν, να βρεθούν συνέργειες μεταξύ των δύο αυτών προσεγγίσεων. Και πολιτικώς το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει. Στις τελευταίες τρεις ε, διασκέψεις που έλαβαν χώρα για το θέμα αυτό, η συμμετοχή ε, είναι όλο και πιο ευρεία. Όλα τα κράτη-μέλη εκτός από ένα παραβρέθηκαν, όπως σας είπα, στη Βιέννη μετά από τη συνάντηση στον aid υπήρχε σαφής ε, αντίληψη ότι κάποιοι είχαν περιθεροποιηθεί στις συζητήσεις και ότι δεν ήταν ικανοποιημένοι με τα πορίσματα των συζητήσεων. Αλλά μετά τη Βιέννη, βάση περιπτώσει, φαίνεται υπάρχει, ότι υπάρχει ένα συγκερασμό των δύο αυτών στρατοπέδων. Και πιστεύω ότι παρά το γεγονός ότι πολλές κυβερνήσεις θα επιλέξουν την βαθμιαία προσέγγιση, βήμα προς βήμα, αυτή η συζήτηση για τον ανθρωπιστικό αντικτύπο έχει ανανεώσει με μεγάλο σημαντικά την όλη συζήτηση. 25 χρόνια συζητάω τα θέματα αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια αίσθηση ανανέωσης, μπορούμε να το πούμε αυτό. Θα πρέπει να αντιτηρηθεί λοιπόν η πίεση θα πρέπει να αποφύγουμε να σκεφτόμαστε υπό τους όρους δύο αντιμαχόμενων, αντίπαλων στρατοπέδων. Θα το συνεχίσει αυτό η Μιρεμπέκα, είμαι σίγουρος. Δεύτερο ζήτημα. Ο αφοπλισμός ως ιδεολογία. Ό,τι και να πιστεύουμε για τις δύο προσεγγίσεις αυτές, σκεφτόμενοι τις ε, συνθήκες για την ε, Συμφωνία Μη και όλες τις σχετικές διασκέψεις, Αν δεν υπάρχει σημαντική πρόοδος τουλάχιστον στον πυρηνικό αφοπλισμό που να είναι ορατή και να προβάλλεται και μία επαναδέσμευση για το σχέδιο δράσης και επαναχωρήσουμε σε σχέση με το σχέδιο δράση, είναι σαφές ότι πέρα από την πολιτική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλέ από τι συμφωνίε αυτέ θα αρχίσουν να αποδυναμώνονται. Πολλά κράτη-μέλη δεν πιστεύουν ότι είναι απλά αυτά. Άρα, στην συνθήκη εξ αρχή ορίζεται ότι χωρίς ε, ορατή δέσμευση για τον πυρηνικό αφοπλισμό το καθεστώς αυτό θα αρχίσει να καταραίει και να μπαίνει σε δύσκολες ε, περιόδους σε σχέση με αυτά που είπε και ο κύριος Walker περιλαμβάνει και περιγράφει τα πυρηνικά στη στρατηγική του σφαίρα όπως η Ρωσία και ύστερα στην ε, χρήση σε ό,τι τη μη διάδοση. Αν αληθεύει λοιπόν αυτό, θα μπούμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Τρίτο θέμα, πυρηνική ασφάλεια και συνεργασία. Πώς μπορούμε να κοιτάξουμε και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα μη διάδοση και ποιοι κίνδυνοι εμπλέκονται. Ω τώρα, σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και μέχρι πριν από κάποιου μήνε, μέχρι τα τέλη του περασμένου έτου, υπήρχε μια σιωπηρή συμφωνία μεταξύ ΙΠΑ και Ρωσία να μην αγγίξουν τη συνεργασία για τη μη διάδοση και για πολλά θέματα, ανεξάρτητα με τις διαφορές που υπήρχαν για την Ουκρανία. Η αντίληψη ήταν ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφέρον να συνεργάζονται για την μη διάδοση περνικών όπλων. Η Συρία αποτέλεσε το πρώτο παράδειγμα χώρας στην οποία συνεχίζονταν η συνεργασία. Υπήρξε ανακοίνωση της Ρωσίας να μην συμμετάχει να συμμετάσχει στην διάσκεψη ασφαλείας του 2016. Αλλά πέρα από αυτό, τα πιο πολλά προγράμματα συνεχίστηκαν. Αυτό μάλλον αλλάζει. Πολύ φοβάμαι και ελπίζω να κάνω λάθος. Η Ρωσία τερματίζει τέτοια προγράμματα στη Ρωσία για να εξασφαλίσει πυρηνικό υλικό. Κι αν λοιπόν επηρεαστεί αυτή η πτυχή της συνεργασίας, αυτό θα έχει αρνητικά αποτελέσματα για όλους μας και θα μπορούσε να επιδεινωθεί πολύ περαιτέρω η κατάσταση. Γίνεται λοιπόν μια συζήτηση για τη συμφωνία και ό,τι και να γίνει στην ε, Ευρώπη. Θα πρέπει να θεωρούμε προς το συμφέρον μας τη συνέχιση τέτοιων συνθήκων. Υπάρχει λοιπόν πραγματικός κίνδυνος σε ό,τι αφορά τις συνέπειες ε, της κρίσης που ενδεχομένω να καταλύσουν και προηγούμενες συμφωνίες. Θα πρέπει σίγουρα να το κοιτάξουμε αυτό. Κοιτώντας όμως τι αποτρέπουν αυτές τις συμφωνίες την πιθανότητα εκ νέου ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι προ το συμφέρον κανενό, προφανώ. Εδώ έχει να διδραματίσει ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ ασχολείται με πιο πολλά στρατιωτικά ζητήματα για την ανάπτυξη ε, όπλων ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα έχει μία φωνή η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά και τη διατήρηση των συνθήκων που ήδη υπάρχουν και την ενίσχυση και την διατήρηση της συνεργασίας που υπάρχει και την πρόληψη α, της διάδοσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το παρελθόν έχει χρηματοδοτήσει και πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες και αυτό παίζει το ρόλο του στη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε τρόπους να προωθηθεί αυτή η συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Ο Ντίτα σου έχει Σας ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Και ευχαριστώ και όλου σα θερμά για τις πολύ εύστοχες ερωτήσεις που εμπλουτίζουν και δίνουν τροφή στη συζήτηση. Κύριε Σαβάιος, συμφωνώ σε πολλά σημεία μαζί σας. Μιλήσατε για την ανθρωπιστική διάσταση που θα πρέπει να συνδυαστεί όχι μόνο με τη συζήτηση της ε, ανάγκης του πυρηνικού αφοβλισμού, αλλά και τη συζήτηση για την πυρηνική ασφάλεια. Συμφωνώ. Είναι ένα θέμα της πυρηνικής ασφάλειας, το ανθρωπιστικό, που δεν ε, ε, εξετάζεται στις διασκέψεις κορυφής για την πυρηνική ασφάλεια. Οι διασκέψεις αυτέ μιλούν για πρόληψη, για λαθρεμπόριο πυρηνικού υλικού, για την πυρηνική τρομοκρατία και αμελούν το ανθρωπιστικό θέμα. Θα πρέπει όμω να είμαστε ρεαλιστέ να δούμε πώ ε, και από πότε και από ποιον μπορεί ένας τρομοκράτης να προμηθευτεί τέτοια πυρηνικά υλικά για να φτιάξει μια βρώμικη βόμβα ή θεός φυλάξη να φτιάξει ακόμη και πυρηνικό όπλο. Είναι πολύ περίπλοκη η ανείχνευση και η κατασκευή τέτοιων πραγμάτων γίνεται μέσω κλοπών τέτοιων υλικών ή μέσω τη ε, μαύρη αγοράς του ελαφρεμπορίου τέτοιων πυρηνικών όπλων. Εννέα χώρε μόνο στον κόσμο έχουν πυρηνικό πλωστάσιο. Από αυτές λοιπόν προέρχονται αυτά τα ε, υλικά και το δικό τους πυρηνικό πλωστάσιο, οι δικέ τους πυρηνικέ κεφαλές ε, δημιουργούν τον κίνδυνο και τι απειλέ στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέρονται πυρηνικές κεφαλές σε κανονικούς οδικούς άξονες από τον χώρο κατασκευής τους μεταφέρονται στην Σκοτία και αποθηκεύονται και, και μεταφέρονται σε αμερικανικούς πυράβλους ή σε πυρηνικά υποβρύχια. Κάθε λοιπόν χώρα που έχει πυρηνικό πλωστάσιο δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας ε, και μία πιθανή πυρηνική απειλή. Και αυτά συζητήθηκαν και στις τρεις ε, διασκέψεις, Όσλο, Ναϊάρτ, Βιέννης και στην επόμενη φαντάζομαι. Είναι ένα τμήμα του, της πολύμορφης συζήτησης και της πολύπτυχης συζήτησης ε, που γίνεται. Και όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία δημιούργησαν το κινητήριο μοχλό για την ε, συνθήκη περί Και είναι εκνευριστικό που μερικές φορές ε, κάποια επιχειρήματα για την ανθρωπιστική διάσταση δεν έχουν ε, την ίδια βαρύτητα με τα υπόλοιπα επιχειρήματα της δημιουργίας των πυρηνικού προστασίου και των επιμέρους θεμάτων. Και κακώς. Το θέμα είναι Ποια στοιχεία λαμβάνονται υπόψη στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Τώρα βρισκόμαστε το 2015 και με ποιο τρόπο θα πρέπει να, να παραταχθούν αυτά τα στοιχεία το ένα δίπλα στο άλλο για να δημιουργηθεί μια δεδομένη ορμή. Η συνθήκη περί μη διάδοση των πυρηνικών αποτέλεσε σημαντικότατο ακρογωνιαίο λίθο για όλους τους στόχους και για όλο το έργο μας ε, υπέρ της αποπυρηνικοποίησης, του πυρηνικού αφοπλισμού και της ε, Πυρηνική ασφάλειας. Δυστυχώς διαβρώνεται η συνθήκη αυτή για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν εφαρμόζεται ο πυρηνικό εφοπλισμός και αυτός είναι ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους ε, οι χώρες χωρίς πυρηνικά αρχίζουν και χάνουν την ελπίδα τους για την αποτελεσματικότητα της συνθήκης αυτής. Ο πρόεδρος Ομπάμα, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησαν σε άλλους τομείς να συνάψουν ε, συμπληρωματικές συμφωνίες, είτε ad hoc συμφωνίες είτε συνθήκες. Και όπως είπα προηγουμένως, το γεγονός είναι ότι πολλές πυρηνικές χώρες είναι κατά της ε, συνολικής συμφωνίας για την ολοσχερή απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Θα πρέπει όμως να γίνει ένας παραλληλισμός ε, αυτών των δύο σημαντικών συνθήκων, τη NTP και τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, γιατί μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία της ε, συνθήκης ε, για τη μη διάδοση. Τώρα έχουμε και το θέμα το ανθρωπιστικό. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί είναι σημαντικό θέμα πρόοδο, όπω και η συνθήκη την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Αυτά είναι τα επιμέρου στοιχεία που θα βοηθήσει την κοινότητα τη συνθήκη περί διάδοσης αλλά και τι τέσσερι πυρηνικέ χώρε που δεν ε, έχουν προσυπογράψει την NTP ή επειδή χρειάζονται κάποιες ε, πρωτοπολογίες ε, και επειδή δεν είχαν υπογράψει όσο δεν ήταν ε, πυρηνικές χώρες και τώρα που είναι χρειάζεται αυτή η αναθεώρηση, είναι περίπλοκα τα πράγματα, θα πρέπει όμως να δούμε το θέμα. Έχουμε το Πακιστάν, τη Βόρεια Κορέα που είναι εκτός του NTP. Και υπάρχει και αυξανόμενη πίεση για την εφαρμογή του άρθρου 6. Μία τέτοια συνθήκη λοιπόν θα αυξήσει και θα ασκήσει πίεση για τις υποχρεώσεις ε, του άρθρου 6. Με τη συνθήκη για την απαγόρευση των ε, πυρηνικών ε, δοκιμών δεν κατα... κατάργησε την ανάγκη εφαρμογή του άρθρου 6 του NTP. Απλώς κάτι που απογορευόταν στην αρχική MPT, δηλαδή οι πυρηνικές δοκιμές για πολιτικούς στόχου τώρα απαγορεύεται. Θα πρέπει επίση να βρούμε τον παραλληλισμό μεταξύ των δύο συνθήκων είναι σημαντικά δομικά υλικά και οι δύο συνθήκε. Επίσης θα πρέπει και οι χώρες που δεν έχουν πυρηνικά να συμβάλλουν στην όλη συζήτηση. Γιατί και αυτές οι χώρες έχουν υποχρεώσει, δυνάμει τη NTP για πυρηνικό αποπλισμό. Επαναλαμβάνω, η υποχρέωση πυρηνικοποίηση δεν αφορά μόνο τις χώρες που έχουν πυρηνικά. Η ε, κυρία Γιάλα με ρώτησε πώ γίνεται αυτό ο αφοπλισμός, η αχρήστευση του πυρηνικού οπλοστασίου. Έχετε δίκιο, το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό ή στρατιωτικό. Παρόλο που και αυτά τα σκέλη είναι πολύ σημαντικά και το τεχνικό και το στρατιωτικό. Αλλά υπάρχει και μια σημαντική πολιτική και κοινωνική πτυχή. Είναι και πολιτικέ και κοινωνικέ διαδικασίε. Εγώ έχω σπουδάσει πυρηνική φυσική. Η τεχνική και η στρατιωτική πτυχή είναι πολύ σημαντικέ ε, και πολύ δύσκολε. Αλλά χρειάζονται ε, και το είδαμε και στην περίπτωση των χημικών όπλων πόσο δύσκολη είναι η τεχνική και η στρατιωτική φάση του παροπλισμού. Από πυρηνική άποψη όμως εξαιτίας της MTP το βασικό έργο της ε, αχρήστευσης των πυρηνικών ε, θα πρέπει να γίνει μόνο από τις χώρες που έχουν τα πυρηνικά. Και αυτό γίνεται με αμοιβαίο έλεγχο. Πάντω ο ρόλο των χωρών που δεν έχουν πυρηνικά και θα θέλω να, να αποτίσω φόρο τιμή ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί χρησιμοποίησε, ε, και στις ε, διαβουλεύσεις στην κοινωνία των πολιτών ε, θα πρέπει και οι χώρες που δεν διαθέτουν πυρηνικά να είναι σίγουρες ότι όντω λαμβάνει η χώρα από πυρηνικοποίηση των χωρών που έχουν τα πυρηνικά. Επίσης, έχουμε στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασιλείο και σε άλλες εννέα χώρες εργαστήρια πυρηνικών. Η, ο, ο παραπλησμός των πυρηνικών κεφαλών είναι γνωστός πώς γίνεται. Αλλά τώρα για να χρησιμοποιηθούν τα επιμέρους υλικά και να ε, χρησιμοποιηθούν το πλουτόνιο και το εμπλουτισμένο ουράνιο για να χρησιμοποιηθούν τα υλικά της επόμενης γενιάς, τα πυρηνικά όπλα της επόμενης γενιάς και ο εξυγχρονισμός του πυρηνικού προστασίου. Αυτό είναι ένας από τους κινητήριους μοχλούς για τη διάβρωση της αξιοπιστίας του NPT για πολλές άλλες χώρες. Γιατί βλέπουν ότι όχι μόνο δεν γίνεται από πυρηνικοποίηση, αλλά εξυγχρονίζεται το πυρηνικό πλωστάσιο των χωρών. Και όποιο σκοπό και αν έχουν ε, ε, οι πυρηνικές, ε, το πυρηνικό πλωστάσιο, κάθε ηγέτης επικαλείται άλλους στόχους, το θέμα είναι ότι περάσαμε από τη φάση της αποτροπής ε, και της τελικής διαβεβαίωσης ε, σε, σε άλλη φάση, γιατί περισσότερες χώρες έχουν το θέμα της αποτροπής. Αλλά εδώ έχουμε μια σχέση μεταξύ των πιθανών αντιπάλων και εξαρτάται από μία σειρά στρατητικών και μη στρατητικών εργαλείων και δεν είναι κάτι που αφορά συγκεκριμένο πυρηνικό όπλο. Νομίζω ότι είναι λάθο και παρεξήγηση τη αποτροπή αν θεωρούμε ότι η αποτροπή εξασφαλίζεται μόνο με την κατοχή πυρηνικών όπλων. Πάντως ακριβώς επειδή δόθηκε στα πυρηνικά όπλα αξία αποτροπής πολεμική σε πολλές χώρες αυτό συνέβη τη πολιτική του επικράτησε σε πολλέ χώρε και μερικέ φορέ και μέσα των Ηνωμένων Εθνών. Θα πρέπει όμω ε, να μειώσουμε τα πυρηνικά και σταδιακά να περάσουμε στην αποπυρηνικοποίηση. Και θα πρέπει να πιέσουμε όλες τις χώρες που έχουν πυρηνικά να μειώσουν και ταυτόχρονα να μην εξυγχρονίσουν το πυρηνικό τους σε επίσης ε, να παροπλήσουν και να διαθέσουν με ασφάλεια τα επιμέρους στοιχεία των πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια συνθήκη που θα απαγορεύει τη χρήση, ανάπτυξη, αποθήκευση, παραγωγή, μεταφορά, διάδοση πυρηνικών ή και τις επιχειρησιακές συναφείς δραστηριότητες που, σχέση έχουν, έχουν σχέση με την προετοιμασία της χρήσης των πυρηνικών και να απαιτήσουμε την ολοσχερή τους ε, κατάργηση. Και γι' αυτό λέω ότι αυτή η συνθήκη είναι το βήμα για μια επόμενη συνθήκη, μια συνθήκη που θα εφαρμόζουν και οι χώρες που δεν έχουν πυρηνικά, ακόμη και αν οι χώρες με τα πυρηνικά αρχικά ε, είναι κατά όπως συνέβη με το CTBT, με τις α, α, ε, νάρκες, ξηράς και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που θα τεθεί σε εφαρμογή μια τέτοια συνθήκη θα αλλάξει πλήρως το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται οι χώρες με τα πυρηνικά, γιατί θα αυξηθούν οι πιέσεις προς αυτές να εφαρμόσουν το άρθρο 6 και οι χώρες εκτός MPT θα αισθανθούν την πίεση και την ανάγκη πυρηνικού αφοπλισμού. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μόνο θέμα εξακρίβωση των τεχνικών ε, θεμάτων σε αυτό το σε αυτό το στάδιο, γιατί αυτά είναι περίπλοκα θέματα και θα πρέπει να τα αναλάβουν οι χώρε με τα πυρηνικά. Αν του περιμένουμε όμω αυτές να συμφωνήσουν μεταξύ τους, ζήσε μου. Φανταστείτε να περιμένουμε από τη Συρία να παροπλήσει όλα τις, τα χημικά όπλα πριν διαπραγματευτούμε και εφαρμόσουμε τη συνθήκη για τα χημικά όπλα. Δεν θα είχε, είχαμε κανένα ε, αποτέλεσμα. Η πραγματικότητα όμως ε, μιλάει για κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να αλλάξει το καθεστώς του όπλου, να απαγορευτεί και μετά να δούμε πώς, ε, τι θα κάνουμε για να απαγορευτεί και να έχουμε και ένα χρονοδιάγραμμα για τον παροπλισμό. Όλα αυτά γίνονται με διαπραγματεύσεις και τότε η συνθήκη γίνεται ο βασικός πολιτικός κινητήριος μοχλός για να αλλάξει και η νοοτροπία των χωρών. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Παρακαλώ ολοκληρώστε. Σας ευχαριστώ, λέει η Κυρία Γκάνσλαντ, ζήτησε το λόγο και ο Μάρκ Γιούρεκ μετά από εσά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές εδώ. Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια. Η σημαντική αυτή ευκαιρία εδώ να τονίσουμε τη σημασία της διάσκεψης αναθεώρησης ε, της συμφωνίας NPT και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε. Τόνισα εξ αρχής ότι η διάσκεψη αναθεώρησης NPT είναι πάρα πολύ σημαντική. Γεγονός κλειδί για μας σε ό,τι αφορά το θέμα της δοφοπλισμού. Και φέτος θα πρέπει να εστιαστούμε για να κάνουμε την διάσκεψη αναθεώρησης μια επιτυχία. Να σας αναφέρω συγκεκριμένα ότι από πλευρά της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θα συνεχίσουμε να διαβουλευόμαστε με εταίρους από όλο τον κόσμο και νομίζω ότι αξίζει να αναφέρουμε ότι για παράδειγμα καλέσαμε τον ε, πρόεδρο τη Αλγερίας, πρέσβη Φαρουκή, να έρθει στι Βρυξέλλε και να μιλήσει στη συζήτηση για την μη διάδοση το Δεκέμβριο. Αυτό καταδεικνύει τις προσπάθειες που κάνουμε να ακούσουμε όλους τους εμπλεκόμενου φορείς και να κατανοήσουμε τα ζητήματα που εμπλέκονται. Μία ερώτηση ακούσαμε. Από την κυρία Γιάλα. Αν τα κατάλαβα, τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να βελτιώσει την ορατότητα, την προβολή και να συμβάλλει στη μη περαιτέρω εξάπλωση τέτοιων όπλων μαζικής καταστροφής. Ένα συγκεκριμένο θέμα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να καταστεί επιτυχής η διάσκεψη. Όποτε έχετε επαφές λοιπόν με τρίτες χώρες, ε, είναι ομολογούσα από χώρες NPT, θα πρέπει να τονίζετε αυτό το μήνυμα. Το πόσο χρειάζεται να ενισχυθούν τα καθεστώτα μη διάδοσης για να υπάρχει ισόρροπο αποτέλεσμα της διάσκεψης του 2015 και να πετύχουμε την ακτή αυτή πρόοδο που όλοι επιθυμούμε σε ό,τι αφορά για τους στόχους που κατοχυρώνονται στην ΠΤ. Αυτό αφενός αφετέρου κάτι διαφορετικό. Να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενεργή για να προωθήσει μέσω συγκεκριμένων έργων τις αρχές που έχουμε, τις πολιτικές αρχές που έχουμε για τον αφοπλισμό. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν χρηματοδοτούμε μία σειρά συγκεκριμένων έργων και υποστηρίζουμε την διεθνή η υπηρεσία ατομική ενέργειας, τη συνεκτική, τη CDBTO. Ως παράδειγμα να αναφέρω εδώ ότι από το 2006, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δαπανίσει 50 δις ευρώ για την υποστήριξη του CBT Όλα αυτά τα παραδείγματα αποτελούν πρακτική, πρακτικά παραδείγματα υποστήριξης στρατηγικής και θα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Χαιρόμαστε για την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ενδεχομένω να υπάρχουν και επίπροσποτετές ερωτήσεις, αλλά υποσχέθηκα στο Μάρεκ Γιούρεκ ε, το λόγο, αλλά έχουμε μόνο λίγα λεπτά διερμηνίες ακόμα μπροστά μας. Ευχαριστώ. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπώ μια χώρα που δεν έχει πυρηνικά, αλλά έχει όμορες χώρες με πυρηνικά. Γι' αυτό είμαι υπέρ της μη διάδοσης. Και αυτή η αρχή της μη διάδοσης δεν θα πρέπει να γίνει αντικείμενο χειραγώγησης. Εδώ και 15 χρόνια η Ρωσία εφαρμόζει ένα πολεμικό δόγμα που επιτρέπει εισβολή ε, η επίθεση σε χώρα που δεν έχει πυρηνικά. Μια χώρα με πυρηνικά ασκεί επίθεση σε χώρα που δεν έχει πυρηνικά. Και το memorandum που ήταν ουσιαστικά η εφαρμογή της αρχής για τη μη διάδοση ε, υπεγράφει μεν αλλά καταπατήθηκε φέτος. Και οι Ινστιτούτα όπως ε, της κυρίας Τζόνσον που δραστηριοποιούνται για αυτά τα θέματα της μη διάδεσης ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το γενικότερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, γιατί θα πρέπει να δούμε τα γενικότερα θέματα της παγκόσμιας δημόσιας τάξης και της προστασίας της ασφάλειας και όχι μόνο να επικεντρωθείτε σε αμυγός τεχνικά ζητήματα Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσετε απαραίτητα. Έτσι, μία σας παρακαλώ. Ναι, είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα θέματα αυτά. Όλα τα θεσμικά όργανα σε σχέση με την αφοπλισμό και την ασφάλεια θα πρέπει να έχουν τεχνικά στοιχεία, τεχνικές ικανότητες. Θα πρέπει όμως να επηρεάσουν και την πολιτική συμπεριφορά. Αυτό που λέμε είναι ότι τα βήματα αυτά θα πρέπει να υπάρχει ο πιο επικοδομητικός διάλογος που γίνεται για το πιο σωστό αποτέλεσμα προκειμένου να έχουμε καλύτερα εργαλεία τελικά να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα προβλήματα αυτά τα οποία τονίζεται. Όπου τα κράτη με πρινικά όπλα δεν συνάδουν με, και δεν συμμορφώνονται με τις εξελίξεις και με τους νόμους και σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που ανακύπτουν από τα πρινικά όπλα. Ελπίζω λοιπόν να υποστηρίξετε μια πρωτοβουλία όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα καταρτήσει ένα ψήφισμα και θα εκφράσει την ομόνια του για θέματα όπως ο ανθρωπιστικός αντικτύπος και για βασικά ζητήματα το πώς αυτό θα προωθήσει όχι μόνο τον αφοπλισμό αλλά και την ασφάλεια και τη μη διάδοση. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που πρέπει να διακόψουμε. Θα ήθελα να έχουμε την ευκαιρία να πούμε πόσο ευγνώμονες είμαστε για τους διερμηνείς μα, τους διερμηνείς μας για τον επιπλέον χρόνο που μας έδωσαν για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.